Καλημέρα και καλώς ήρθατε όλοι σας. Ξεκινάμε με την έγκριση της ημερησίας διατάξεως. Όπως σας ενημέρωσε η γραμματεία, θα υπάρξει μια πρωτοβουλία ή μια ε, αποτελεσματική ε, εταιρική ε, συνεργασία. Θα λάβει χώρα αύριο στις 11 και όχι το απόγευμα. Επίσης, για την έχουμε προβλέψει για το πρωί της Τρίτης για το Mercosur και σας ενημερώνω ότι οι συζητήσεις ε, συνεχίζονται στην ομάδα εργασίας. Γι' αυτό σκεφτήκαμε ότι θα ήταν πρόωρο να παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα της ομάδας εργασίας. Επίσης, προσθέθηκε ένα επιπλέον θέμα από την ε, Επιτροπή Αλίας για την εταιρική σχέση Ευρωπαϊκή Ένωση με τα νησιά του Σάλωμο όπου θα έχουμε και εισηγητή. Δεν ξέρω αν υπάρχουν κάποιες ε, επιφυλάξεις όσον αφορά την ημερήσια διάταξη, όπως έχει. Άρα μπορώ να θεωρήσω ότι εγκρίθηκε. Επίσης, έχετε τα πρακτικά τη 26-27 Απριλίου του 2010. Αν έχετε κάποιε παρατήρησει να κάνετε πάνω σε αυτά τα πρακτικά, να το πράξετε στη γραμματεία μέχρι το, πριν να τελειώσει η συνεδρίασή μα. Ε, θα θεωρήσουμε ότι έχουν εγκριθεί. Ανακοινώσεις Προέδρου δεν υπάρχουν. Τώρα μήπως έχει κάποιε ανακοινώσει να κάνει η Επιτροπή. Όχι. Λοιπόν, δεν έχουμε κανένα ερώτημα να θέσουμε στην Επιτροπή. Εγώ προσωπικά που έχω προβλέψει κάποια ερώτηση θα το δούμε τον Ιούλιο. Άρα, Πηγαίνουμε στο σημείο 6. Τροποποίηση του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση μηχανισμού χρηματοδότηση τη αναπτυξιακή συνεργασία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λοιπόν, ε, για το θέμα της συμφωνίας ε, για την μπανάνα, ένα θέμα το οποίο έχει διαμαρτυρηθεί η Ευρώπη, έχει δημιουργηθεί ένα πρόγραμμα για να παρακολουθήσει το θέμα του χώρου αυτού στις χώρες ΑΚΕ ε, που προμηθεύουν, ε, παράγουν τέλο πάντων μπανάνε. Έχουμε την έκθεση του κύριου Γκέρενς και οι σοντινσές θεωρούν ότι χρειάζεται η γνωμοδότηση ενός εξωτερικού εμπειρογνώμονα να γίνει μια ανάλυση σε βάθος για τα κεφάλαια και τα φρούτα αυτά και Υπάρχει πρόθεση σε σχέση με το εμπόριο της μπανάνας στην Λατινική Αμερική, στην Καραϊβική και τους προορισμούς που αφορούν την ευρωπαϊκή αγορά. Θα δώσουμε το λόγο στο Σιγβίντ, ειδικό εμπειρογνώμων του Ινστιτούτου. Θα δώσουμε το λόγο, εκπροσωπείται μάλλον από τον κύριο Μαραζάν και θα του δώσουμε τώρα το λόγο. Θα μιλήσω ισπανιστή. Ευχαριστώ πολύ. Για να μπορέσουμε να αναλύσουμε την κατάσταση της αγοράς μπανάνας και τις ενδεχόμενες ε, συνέπειες που θα προκύψουν από τη Συμφωνία της Γενέδης θα ήθελα καταρχήν να σας δώσω μια γενική επισκόψη τη ιστορική κατάσταση της αγοράς μπανάνας που βλέπετε σε αυτό το γράφημα Πάνω από 60% των εισαγωγών μπανάνα πηγαίνουν στι Ηνωμένε Πολιτείε και στις Ηνωμένε Πολιτείε. Μεγάλη σημασία έχει φυσικά και η αγορά της ε, πάλι ποτέ Σοβιετικής Ένωσης και χωρών αναπτυσσομένων όπως η Κίνα. Η πολιτική εμπορίου για τις μπανάνες επηρεάζεται στην ευρωπαϊκή αγορά από τρία πάρα πολύ σημαντικά στοιχεία. Πρώτα απ' όλα από τις συμφωνίες Κοτονού, τις συμφωνίες που υπάρχουν λοιπόν με τις χώρες ΑΚΕ, στα πλαίσια των, ε, της ε, συνθήκης Κοτονού και στις εταιρικέ οικονομικές ε, συμφωνίες. Δεύτερον, μέσα στα πλαίσια των κανόνων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, της ρήτρα πλέον ευνοούμενου έθνους και του γύρω της ε, Ντόχα και τέλος στην περίπτωση Λατινικής Αμερικής τις συμφωνίες ε, σύνδεσης που έχουν υπογραφεί ή που επίκειται η υπογραφή τους όπως στην περίπτωση της κοινότητας των Άνδρων που έχουν μια πολύ μεγάλη σημασία σε ό,τι αφορά την ε, κατάληψη της αγοράς σε βάρος των χωρών ΑΚΕ. Αν δούμε τώρα πώς έχει η κατάσταση της ευρωπαϊκής αγοράς σε ό,τι αφορά τις εισαγωγές αναχώρα προέλευσης, βλέπουμε ότι πάνω από το 70% των εισαγωγών μπανάνας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ερχόνται από τη Λατινική Αμερική, <clears throat> ιδίως από το Εκουαδόρ, την Κολόμβια και την Κωνσταντίνα. Και ένα ίσον τμήμα άρχεται από τις χώρες ΑΚΕ. Μέσα στις χώρες αυτές ε, ΑΚΕ, τα δύο τρίτα προέρχονται από το Καμερούν και από την ακτή του Ελεφαντοστού και το τελευταίο τρίτο από τις χώρες Καραϊβικής. Βλέπετε στο γράφημα επίσης την κατανομή μεταξύ των δύο μπλοκ χωρών, αφενός των χωρών της Λατινικής Αμερικής και δεύτερον των χωρών ΑΚΕ. Από το 2006 υπήρξε μια σημαντική αύξηση στις εισαγωγές λόγω της κατάργησης των ποσοστώσεων στις εισαγωγές από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά βλέπετε ότι αυτή η μεταρρύθμιση της αγοράς ουσιαστικά σε μόνο τη Λατινική Αμερική. Τώρα, στην Γενέβη υπήρξε μια συμφωνία στα πλαίσια του ΠΟΕ που προβλέπει μια <clears throat> σταδιακή μείωση των δασμών από 176 δολάρια τον τόνο σε 114 δολάρια για το χρονικό διάστημα 2009 έως 2017. Επίσης, με μια συμφωνία προτιμησιακού χαρακτήρα για τα τροπικά προϊόντα. Γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αποφασίσει να αναλάβει συνοδευτικά μέτρα στην αγορά της μπανάνας που <clears throat> περιλαμβάνουν και μία υποστήριξη 190 εκατομμυρίων δολαρίων για τους παραγωγούς των χωρών ΑΚΕ που θα χάσουν ουσιαστικά το προτιμησιακό τους καθεστώς, θα διαβρωθεί το προτιμησιακό τους καθεστώς βάσει της συνθήκης Κοτονού. Είναι πολλοί οι εμπειρογνώμονες οι οποίοι έχουν κάνει κάποιες προβλέψεις για το τι θα γίνει με την μείωση των δασμών. <clears throat> Στο γράφημα αυτό μπορούμε να δούμε ποια είναι τα δυνητικά σενάρια τα οποία μπορεί να λάβουν χώρα ξεκινώντας από το δασμό των 176 ευρώ που ήταν αρχικά και φτάνοντας στο τελικό επίπεδο του μηδενικού δασμού. Αυτό δείχνει πώς θα τροποποιηθεί η μερίδα αγοράς για τις χώρες με καθεστώς πλέον ευνομούμενου κράτους, που είναι κυρίως οι χώρες της Λατινικής Αμερικής, όσο μειώνονται οι δασμοί, όλο και περισσότερε θα είναι εισαγωγές από τις χώρες αυτές και όλο λιγότερες θα είναι εισαγωγές από τις χώρες ΑΚΕ. Κατά τρόπον ώστε οι συμφωνίες στα πλαίσια του ΠΟΕ θα έχουν ένα πάρα πολύ σημαντικό αρνητικό αντίκτυπο για τις χώρες ΑΚΕ. Επίσης, άλλες προβλέψεις που βασίζονται σε διάφορα επίπεδα δασμών που τα βλέπετε στα αριστερά, με τα 159 ευρώ μέχρι το 0 δείχνουν και την ελαστικότητα της ε, καμπύλης προσφοράς από τις χώρες της ε, Καραϊβικής. Η Τσαμάικα, παραδείγματος χάρη, θα χάσει πάνω από το μισό των εξαγωγών της αν φτάσουν οι δασμοί στο μηδέν και αυτή είναι η γενική κατάσταση των χωρών της Καραϊβικής. Είναι οι χώρες οι οποίες θα θυγούν περισσότερο από την φιλελευθερωποίηση του εμπορίου της μπανάνας. Τι σημαίνει αυτό σε ό,τι αφορά την αλυσίδα προσθέμενης αξίας <laughs> στην αγορά της μπανάνας. Αυτό το οποίο θέλω να τονίσω καταρχήν είναι ότι δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή εκτιμήσεις οι οποίες να είναι εμπεριστατωμένες. Υπάρχουν στοιχεία διάσπατα και πληροφορίες διαφόρου χαρακτήρα που έχουν συλλεγεί από διάφορους φορείς, αλλά έχουν ένα χαρακτήρα απόλυτα αποσπασματικό. Εδώ έχουμε τα στοιχεία της αγγλικής ε, International Food Group <clears throat> και λέει ότι αν πάρουμε ένα κιλό μπανάνας, το 40% των κερδών από, τα, από το ένα κιλό αυτό μπανάνας θα πάνε στα υπερκαταστήματα, στους λιανοπολιτές, το 17% στους διανομείς και το 31 έως 36% στις εταιρείες οι οποίες εμπορεύονται το, τις μπανάνες, η τσικίτα, ντόλε και ντελμόντε. Αλλά στη χώρα προέλευσης παραμένει μόνο το 11,5 της συνολικής αξίας, από το οποίο 1,5 αφορά την αμοιβή των εργαζομένων στις φυτίες μπανάνας. <clears throat> Αυτή είναι μια κατάσταση η οποία ισχύει όχι μόνο για τους παραγωγικούς μπανάνας στις χώρες της Αμερικής, αλλά και για πολλούς παραγωγούς μπανάνας που εξάγουν προς την Ευρώπη όπως είναι το Καμερούν ή η ακτή ελεφαντοστού. Η μόνη διαφοροποίηση είναι οι περιπτώσεις των ε, προσύνεμων νήσων στις Καραϊβικές, στην Καραϊβική όπου οι μικροί παραγωγοί μπορούν να έχουν πολύ μεγαλύτερα ποσοστά ε, προσθέμενης Στα πλαίσια του εμπορίου της μπανάνας μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν δύο υποδείγματα για την αλυσίδα προσθέμενης αξίας που επικρατούν αυτή τη στιγμή. Με τρεις κρίκους. <clears throat> Στον πρώτο κρίκο είναι ο άμεσος παραγωγός. Στο δεύτερο κρίκο έχουμε μια ολοκληρωμένη αλυσίδα, η εταιρεία η οποία εμπορεύεται τα προϊόντα αυτά, η Τσικίτα παραδείγματος χάρη, συγκεντρώνει το έργο της ε, συσκευασίας, εξαγωγής, ορίμανσης και διανομής των ε, μπανανών και τα υπερκαταστήματα απλώς κάνουν το λιανικό εμπόριο. Αυτό το οποίο βλέπουμε λοιπόν στο εμπόριο της Πανάνας είναι ότι μετά από τη δεκαετία του 1990 περάσαμε από μια πολύ περισσότερο ολοκληρωμένη αλυσίδα προσθέμενης αξίες όπου οι δραστηριότητες της ε, ε, φυτίας της ε, μπανάνας έχουν ενσωματωθεί σε αυτή τη διαδικασία. Και βλέπουμε τώρα ότι έχουν μείνει ουσιαστικά δύο μονάχα κομμάτια, δύο κρίκες στην αλυσίδα που είναι αυτά που κάνει η εταιρεία μπανάνας και οι λιανοπολιτές. Υπάρχει και το λεγόμενο δίκαιο εμπόριο, το fair trade, όπου γίνεται μια προσπάθεια οι παραγωγοί να έχουν περισσότερα ωφέλη από την δραστηριότητα αυτή της καλλιέργειας, της συσκευασία και της εξαγωγής μπανανών. Αν δούμε ποιε είναι οι αναλύσεις της ΦΑΟ από τα Ηνωμένα Έθνη σε ό,τι αφορά την ε, παραγωγή μπανάνας, Έχουμε κάποια ενδιαφέροντα προϊόντα, εάν αναλύσουμε την αμερικανική αγορά. Την αγορά των ΗΠΑ λοιπόν και της Ευρώπης και εάν αναλύσουμε το πώς κατανέμεται το κέρδος σε αυτή την αλυσίδα μεταξύ των παραγωγών και των καταναλωτών αφενός και μεταξύ και τις διαφορές που υπάρχουν <clears throat> μεταξύ της συμβατικής αλυσίδας προσθέμενης αξίας για την μπανάνα και τις αλυσίδες που ισχύει για τις βιολογικές μπανάνες. Βλέπετε λοιπόν στο γράφημα αυτό ότι η κατανομή των εσόδων μεταξύ στην Αμερικανική αγορά δείχνει να υπάρχει μια διαφορά μεταξύ των ε, βιολογικών και των συμβατικών μπανανών. Οι συμβατικές έχουν κυρίως από το Εκουαδόρ, από τον Ισημερινό και βιολογικές από το Περού, βλέπει κανείς ότι είναι πολύ πιο μικρό το ποσοστό προσθέμενης αξίας που μένει στη χώρα. Η άσπρη ζώνη που βλέπετε είναι αυτό το οποίο αφορά τους δασμούς εισαγωγής στις ΗΠΑ. Αν συγκρίνουμε αυτό με την Ευρώπη βλέπουμε ότι αυτή η λευκή ζώνη που είναι πολύ μικρή είναι το περιθώριο εισαγωγής είναι πολύ πιο μεγάλο στην Ευρώπη. Αυτή η διαφορά λοιπόν καθορίζεται από τους δασμούς που μπορούν να επιτευχθούν. Η τιμή της μπανάνας λοιπόν στην Ευρώπη είναι 130% υψηλότερη από τη τιμή της μπανάνας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Παρ' όλα αυτά, το μεγαλύτερο ποσοστό από αυτής της τιμής, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΦΑΟ που βλέπουμε τώρα, αφορά το κόστος εισαγωγής λόγω των δασμών που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή η διαφορά λοιπόν δεν υπάρχουν για τις ε, βιολογικές μπανάνες που προέρχονται από τη δημοκρατία, Δομινικανική Δημοκρατία που είναι μια χώρα ακέα. Το σημαντικό εδώ που θέλουμε να κατανοήσουμε είναι ότι το σκούρο κομμάτι στο, κάτω μέρος της στήλη δείχνει ότι η διαφορά μεταξύ μιας βιολογικής μπανάνας και μιας κανονικής μπανάνας σε ό,τι αφορά το κόστος παραγωγής και όλα αυτά είναι ελάχιστη. Είναι σημαντικό λοιπόν να δούμε στην περίπτωση της Γερμανίας, ποιο είναι το ποσοστό, ποιο είναι το περιθώριο που μπορούν να, να αποκτήσουν οι εισαγωγείς για τις ε, μπανάνες. Αυτά που είναι το περιθώριο της βιολογικής μπανάνας είναι πιο ψηλό, αλλά τα κέρδη από αυτό δεν μετακυλίζονται στους παραγωγούς. Τέλος, υπάρχει μια διαφορά μεταξύ των διαφορετικών ειδών μπανάνας που την χάνουν εξαγωγής προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε στα αριστερά την συμβατική μπανάνα, στο κέντρο την βιολογική μπανάνα και στα δεξιά τη λεγόμενη μπανάνα fair trade, δικαίου εμπόριου. Αυτό που είναι σημαντικό σε ό,τι αφορά την πολιτική εμπορίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το πιο σημαντικό είναι η πρώτη στήλη, όπου το έσοδο του, εισαγω... του παραγωγού είναι πολύ μικρότερο από ότι αυτό του fair trade. Αλλά αν δούμε τις μπανάνες fair trade που εισάγονται στο Ηνωμένο Βασίλειο από την Καραϊβική βλέπουμε ότι τα κέρδη των ε, υπερκαταστημάτων είναι πολύ μεγαλύτερα από αυτά τα οποία μπορούν να πάρουν από τη σημαντική μπανάνα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν ότι και από τη βιολογική και την κανονική μπανάνα οι μπανάνες fair trade αποκομίσουν περισσότερο κέρδος στα υπερκαταστήματα. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις λοιπόν <clears throat> το περιθώριο κέρδους των υπερκαταστημάτων είναι μεταξύ 40 και 48%. Τόσο η ΦΑΟ όσο και άλλοι εμπειρογνώμονες κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι σήμερα μέσα στην αλυσίδα προσθέμενης αξίας τα μεγαλύτερα κέρδη για την μπανάνα δεν καταλήγουν στις εταιρείε μπανάνες, στην Τελμόντε, στην Σικίτα κτλ. Αλλά οι μεγάλες αλυσίδες υπερκαταστημάτων στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ. Από την άποψη αυτή λοιπόν θεωρούμε ότι υπάρχουν διαφοροποιημένοι αντίκτυποι ανάλογα με τη χώρα στην οποία θα υπάρξουν μέτρα φιλελευθερωποίησης στην Δομινικανική Δημοκρατία, Μπελίσε και Σουρινάμ είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα για την ε, εξαγωγή και την ανταγωνιστικότητα, ενώ η Δομίνικα, Σαν Λούσεν και Σαν Ταλουτσία θα έχουν πολύ μεγάλα προβλήματα σε μια φιλελευθεροποιημένη αγορά και ιδίω αν υπάρχει μεγαλύτερο μερίδιο τη αγορά μπανανών fair trade. Μια ανάλυση λοιπόν των συναλλαγών σε μπανάνα δείχνουν ότι οι χώρες καραϊβικές έχουν πολύ λίγες δυνατότητες να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις μεγάλες απώλειες που οφείλονται στη διάβρωση του καθεστώτος προτιμησιακών εισαγωγών. Έχουν πολλά μειονεκτήματα συντηρητικού χαρακτήρα, το έδαφος, το κλίμα κτλ. Θα είναι πολύ δύσκολο λοιπόν οι χώρες αυτές να μπορέσουν να διατηρήσουν την ανταγωνιστικότητα στο... στην παραγωγή μπανάνας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν έχει τέσσερις επιλογές τουλάχιστον είτε να προσπαθήσει να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα της ε, βιομηχανίας μπανάνας στις χώρες αυτές ή να ξεκινήσει μια διαδικασία αντικατάστασης της παραγωγής μπανάνας ή να ενισχύσει <clears throat> την αλυσίδα παραγωγής fair trade ή να επιτύχει μεγαλύτερη διαφοροποίηση παραγωγής. Για να γίνει κάτι τέτοιο έχουμε να θέσουμε τα εξή ερωτήματα κατά πόσον οι χώρες οι οποίες είναι πιο ανταγωνιστικές μέσα στην ομάδα των χωρών της Καραϊβικής θα απαιτήσουν πρόσθετη βοήθεια. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί. Μιλάω για το Σουρινάμ και την Πελίζε που έχουν δείξει ότι μπορέσαν να επιβιώσουν μέσα στην αγορά την φιλελευθερωποιημένη. Δεύτερον, αντίθετα χώρες που έχουν σχετικά μικρή εξάρτηση από την αγορά μπανάνας όπως η Τζαμάικα που έχουν διαφοροποιήσει την παραγωγή τους ή έχει καταστραφεί η παραγωγή τους. Ποια είναι η καλύτερη δυνατότητα για να ε, υποστηρίξουμε τα προσύνεμα, τις προσύνεμες νήσους και με ποιο τρόπο μπορούμε να έχουμε καλύτερες πληροφορίες για τη διάβρωση του προτιμησιακού καθεστώτος και μήπως θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τα κοινωνικά και οικολογικά πρότυπα για να αποφύγουμε τα αρνητικά αποτελέσματα της διαδικασίας φιλελευθερωπής. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γκέρενς, ο εισηγητής μας έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω καταρχήν το συντάκτη της μελέτης αυτής. Τώρα την ανακαλύπτω, γι' αυτό σας πρότεινα να αλλάξουμε λίγο την μερίσια διάταξη και να του δώσουμε στον κύριο το λόγο να παρουσιάσει το θέμα. Για να διασαφηνίσει το όλο θέμα. Ε, στη διαδρομή που λέω εγώ τη μπανάνας. Εγώ από αυτά καταλαβαίνω ότι καταλαβαίνω ότι από την όλη παραγωγή μόνο 1,5% ότι μένει σαν αμοιβή του, στον παραγωγό. Έχουμε εδώ ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ λεπτό. Είναι παρα, παραπάνω από ένα απλό φρούτο η μπανάνα. Είναι θεσμός θα λέγαμε. Είναι ένας σημαντικός τομέας. Ε, ένα θέμα που είναι, αφορά πάρα πολύ την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σημαντικό τομέα αυτό που έχει να κάνει τι αγωγέ αυτού του φρούτου. Είναι οι χώρε τη ΑΚΕ που, ε, οι οποίε έχουν άμεσο συμφέρον. Απ' την άλλη, είναι προϊόντα τα οποία παράγονται με καθαρό σκοπό τις εξαγωγές. Και αυτό που ίσχυε μέχρι τώρα ήταν και συνεχίζει να ισχύει είναι ένα προτιμησιακό καθεστώς για τις χώρες ΑΚΕ. Στα πλαίσια του ο, ΠΟΕ, εδώ υπάρχει μια, είναι ένα, έχει ένα ιδιαίτερο καθεστώς παρόλο που υπάρχει μια αμφισβήτηση εδώ και 15 χρόνια. Σας υπενθυμίζω ότι υπάρχουν διαπραγματεύσεις όσον αφορά την εμπορική πτυχή, αλλά υπάρχει η πτυχή που έχει να κάνει με την ανάπτυξη. Και είναι σημαντικό αυτό διότι εμεί σαν Επιτροπή ε, αυτό που μας αφορά και αυτός ο οποίος μας ευαίσθη είναι να προωθήσουμε αυτή την πτυχή που έχει να κάνει με την ανάπτυξη. Απ' τη μια έχουμε την αναγκαιότητα σε διεθνές επίπεδο του εμπορίου, απ' την άλλη όμως πρέπει να λάβουμε υπόψη και τα συμφέροντα ε, επιτόπου που έχουν οι παραγωγοί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση σε προήμιο του κειμένου αναφέρει ότι επιμένει στις αρχές της θα πρέπει να συνεχίσουμε να, υποστηρίζουμε τις χώρες ΑΚΕ. Θα γίνει όμως αυτό λίγο λιγότερο τώρα. Οι δασμοί που έχουν να κάνουν με τις μπανάνες που έρχονται από τις άλλες χώρες που δεν ανήκουν στις ε, ΑΚΕ θα έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον και εσείς έχετε περιγράψει τις επιπτώσεις που θα υπάρχουν όσον αφορά την κατάσταση και για το μέλλον αυτής της καταστάσεως. Απ' την άλλη πλευρά φυσικά εμείς είμαστε ρεαλιστές. Διαπιστώνουμε ότι ε, δεν υπάρχουν πολλές ε, ε, εναλλακτικές λύσεις. Απ' τη μια είναι μια συμφωνία στην οποία, η οποία έγινε, για την οποία έγιναν διαπραγματεύσεις, υπήρχε μια πίεση σε αυτήν την κατάσταση. Ε, αναφέρθηκε ότι είχαν ένα προνομισιακό καθεστώς και στο οποίο στην τελική ανάλυση έχει αμφισβητηθεί από τους ανταγωνιστές. Γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ε, αναγκάστηκε να, να αλλάξει την οπτική της γωνία όσον αφορά τις εισαγωγές σε αυτόν τον τομέα. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Δεδομένου ότι όσον αφορά οι, οι εταίροι της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πληρώσουν την κατάσταση αυτή. Ε, έχει προβληθεί εξάλλου μια συμφωνία που έχει να κάνει με αντισταθμίσεις υπάρχει το ποσό των 190 εκατομμυρίων ευρώ και μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση ίσως να μας δώσει λεπτομερείς πάνω σε αυτό. Αναφέρεται περίπου το ποσό των 200 εκατομμυρίων και ενδεχομένως να προσθεθούν άλλα 10 εκατομμύρια για τις χώρες οι οποίες θα πληρώσουν θα λέγαμε όσον αφορά αυτή τη συμφωνία. Αυτή είναι η κατάσταση η οποία χειροτερεύσει σχέση με αυτά που ισχύαν μέχρι πέρσι. Αυτά λέμε ότι είναι συμπληρωματικά μέτρα όσον αφορά την μπανάνα. Ε, ε, υπάρχει το μέσο για την ανάπτυξη και αναφέρεται ότι τα χρήματα αυτά θα χρησιμοποιηθούν για να χρηματοδοτήσουν δράσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την αναπτυξιακή συνεργασία με τις χώρες ΑΚΕ και μπορούμε να πούμε ότι αυτό είναι μια καταρχήν απάντηση προς τις χώρες ΑΚΕ. Μια άλλη πτυχή τώρα που αφορούν τα ε, συμπληρωματικά μέτρα για την μπανάνα. Εδώ έχουμε να κάνουμε με μια ε, στρατηγική που θέλει να υποστηριχθούν οι χώρες οι οποίες θα πληρώσουν για αυτή τη συμφωνία, οι οποίε πλήττονται δηλαδή, και η Επιτροπή θα κάνει διαπραγματεύσεις ε, να πετύχει κάποιες συμφωνίε με αυτές τις χώρες. Σύμφωνα με τι επαφέ που έκανα με την Επιτροπή για αυτή τη συζήτηση, δεν μπορούμε να πετύχουμε μια ε, δεδομένη συμφωνία. Θα υπάρχει διαφορά από χώρα σε χώρα. δεν θα υπάρχει ίδια δηλαδή προσέγγιση για όλες τις χώρες, διότι κάποιες χώρες, για παράδειγμα, έχουν μια διακυβέρνηση που επιτρέπει στην Επιτροπή να προβλέψει ε, ένα, μια συμφωνία στα πλαίσια του προπολογισμού ή τομιακά και με αυτόν τον τρόπο να δώσει ένα μέρος των 190 εκατομμυρίων που προβλέπονται μέχρι το τέλος του 2013. Απ' την άλλη υπάρχουν και χώρες οι οποίες δεν εντάσσονται στο, στην ίδια προσέγγιση αυτή του ανατομέα ή στα πλαίσια του προπολογισμού. Αλλά θα ωφεληθούν μέσω κάποιων προγραμμάτων που θα προγραμματιστούν. Τι μπορούμε να κάνουμε. Έχουμε τη μελέτη που παρουσιάστηκε μόλις τώρα. Να δούμε να, τι μπορούμε να κάνουμε υπέρ των παραγωγών. Να δούμε ποιες είναι οι δυσκολίες και η Επιτροπή μου έδειξε ότι θα είναι δύσκολα. Αυτό μπορεί να γίνει στα πλαίσια του fair trade που αναφέρετε κι εσείς. Ε, ε, ε, είναι μια πολιτική φιλόδοξη και πρέπει να την προωθήσουμε η Επιτροπή θα λάβει η υπόψη λοιπόν τα συμφέροντα των παραγωγών. Προβλέπεται αυτό και είναι κάτι θετικό. Επίσης, αυτό που είναι σημαντικό είναι να υπογραμμίσουμε τη σημασία του να χρηματοδοτήσει κανείς αποκλειστικά με, μέτρα που θα καταπολεμούν την φτώχεια. Αυτός πρέπει να είναι ο στόχος. Να βελτιωθούν οι υποδομές. Επίσης, μπορεί να βοηθήσει ούτως ώστε παραγωγή στις χώρες ΑΚΕ να γίνουν πιο ανταγωνιστικοί. Και όλα αυτά εντάσσονται στα πλαίσια εφαρμογής των συμφωνιών που θα διαπραγματευτεί η Επιτροπή της χώρας αυτές. Δύο έγγραφα λοιπόν, αν κατάλαβα καλά. Ένα που έχει στρατηγική προσέγγιση και ένα άλλο το οποίο θα έχει μια αιτήσια προσέγγιση και το οποίο, τα οποία έγγραφα θα μας υποβληθούν για να τα συζητήσουμε εδώ στην Επιτροπή Ανάπτυξης. Επίσης, αυτό που είναι σημαντικό την εσωμάτωση σταδιακά αυτών των χωρών στην παγκόσμια οικονομία είναι ένα από τους μεγάλους στόχους των ε, εμπορικών συνεργασιών, δαβάνοντας πάντα υπόψη την ανάπτυξη αυτών των χωρών. Χώρες στις οποίες για μεγάλο χρονικό διάστημα ε, προστάτευσε η Ευρώπη, αλλά και εμείς πρέπει να προστατευτούμε, ε, βλέποντας τα πράγματα με μια οπτική που αφορά την παγκόσμια οικονομία. Επίσης κάτι που είναι σημαντικό κατά για, για, μετά το 2013 δεν έχει προβλεφθεί τίποτα. Είναι ενοχλητικό. Τα προγράμματα που δείξατε περισσότερο είναι διαρθρωτικά. Τα διαρθρωτικά προβλήματα λοιπόν δεν θα σταματήσουν όταν θα κλείσει, ε, θα τελειώσουν αυτές οι συμφωνίες. Θα πρέπει λοιπόν η Επιτροπή να προβληματιστεί γιατί το διάστημα μετά το 2013. Ε, γνωρίζω αυτούς, για αυτές τις χώρες. Ε, τα προβλήματα λοιπόν έχουν, είναι διαρθωτικά. Θα πρέπει να δούμε μακροπρόθεσμα το θέμα και να έχουμε μια στρατηγική πιο κατάλληλη να σκύψουμε πάνω αυτό το πρόβλημα. Έχουμε ε, προγράμματα τα ισχύουν για διάστημα 7 ετών, θα πρέπει να δούμε ε, και τις δικές μας ε, συμφέροντα και να δούμε και το χώρο το χωρώνα και Αυτά σαν μια πρώτη αντίδραση σε σχέση με αυτά που μας παρουσίασε ο μιλητής θα πρέπει να δοθεί γνωμοδότηση πάνω σε αυτή τη συμφωνία. Επίσης να πω ότι επιθυμώ να προχωρήσουμε γρήγορα στο έργο αυτό και όσο το δυνατό πιο γρήγορα να έχουμε ένα σχέδιο έκθεσης ούτως ώστε να προχωρήσουμε ούτως ώστε να έχουμε την έγκριση της Επιτροπής. Επίσης έχουν προβάλλει σε όλες τις συζήσεις που κάνουμε με την Επιτροπή ε, το να έχουμε ένα πνεύμα επικοδομητικό και με τη με καλύτερη δυνατή διαφάνεια. Γι' αυτό λοιπόν ζητώ όσο να το πιο γρήγορα να έχουμε ένα σχέδιο συμφωνίας. Αυτό πάνω στο οποίο κάνει διαπραγματεύσει η Επιτροπή με τις χώρες που θα ε, μπορέσουν να έχουν αυτήν τη βοήθεια να γίνει αυτό γρήγορα, ούτω ώστε να προχωρήσουμε. Ε, οδηγούμε λοιπόν σε μια κατάσταση που έχει να κάνει με την κατάργηση του προτιμησιακού καθεστώτος. Αυτά σαν παρατηρήσεις οι οποίες ε, θίγουν τις πτυχές τις πιο ουσιαστικές ε, αυτού του θέματος. Ευχαριστώ, Πρόεδρος. Η κυρία Γκρέσ ζήτησε το λόγο. Ε, Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον ε, κύριο Μοραζάν που μας παρουσίασε την ε, μελέτη του, που στην πράξη επιβεβαιώνει τα όσα είχαμε ήδη διαβλέψει στην στιγμή της υπογραφής ε, των συμφωνιών στις 9 Δεκεμβρίου για την Πανάνα. Άρα λοιπόν τα στοιχεία που μας παρουσιάσατε επιβεβαιώνουν, επικυρώνουν αυτή την ανάλυση και μάλιστα βρήκα ενδιαφέρουσα την ανάλυση σας για το Fair Trade. Είναι αριθμοί, στοιχεία τα οποία εγώ δεν γνώριζα τουλάχιστον. Να ευχαριστήσω επίσης τον κύριο Γκέρενς για την πρώτη του προσέγγιση για την έκθεση που σκοπεύει να κάνει για το θέμα αυτό. Είναι ένα ζήτημα περίπλοκο και πάρα πολύ ευαίσθητο, το οποίο ξεπερνά την, το εμπόριο της μπανάνας. Εγώ ασχολήθηκα και κοίταξα κάπως το περιεχόμενο της πρότασης κανονισμού της ε, Κομισιόν και θα πρέπει να πω πως ήδη έχω πολλά πολλά ερωτήματα. Τονίσατε τρία σημεία. Την ανταγωνιστικότητα, την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, αν μου επιτρέπετε αυτό θα το αφήσω κατά μέρος. Το δεύτερο σημείο είναι η προώθηση της διαφοροποίησης. Εδώ θα ήθελα να επανέλθω. Τα όσα έγιναν σαφή μέσα στην ανάλυση που είδαμε είναι πως όντως το εμπόριο της μπανάνας κυρίως ωφελεί τις μεγάλες επιχειρήσεις και τους μεγάλους, τις μεγάλες εταιρείες δενομής. Και το είδαμε αυτό ότι δηλαδή πολύ λίγα αποφέρει στους μικρούς ε, παραγωγούς και στους ε, εργαζόμενους στον τομέα της μπανάνας. Άρα λοιπόν στα όσα είδαμε για τη διαφοροποίηση υπάρχει μια έκθεση που έχει συνταχθεί για τον τρόπο με τον οποίο έχουν δαπανηθεί τα κονδύλια και διαπιστώνουμε και στην Καραϊβική, αν δούμε ας πούμε το παράδειγμα της Σεντ Λουισί, που ότι δηλαδή ε, δόθηκαν έτσι κατακαιρματισμένα τα κονδύλια αυτά που τελικά δεν είχαν κανένα αποτέλεσμα. Ενώ βλέπουμε ότι για τη διαφοροποίηση τα κονδύλια δαπανήθηκαν σε τομείς που είναι ο τουρισμός, οι υποδομές, η γεωργική ανάπτυξη, ο κατασκευαστικός τομέας και ούτω καθεξής. Ε, και στην επόμενη φάση λοιπόν, και ίσως αυτό θα πρέπει να το συζητήσουμε και με τον κύριο Κέρενς, πάντως ε, η στήριξη στην διαφοροποίηση θα πρέπει να γίνει πολύ πιο στοχευμένα στοχευμένα, ε, δηλαδή κυρίως για τη γεωργία και ίσως ε, και το, στον τουρισμό, αυτό που λέμε στα γαλλικά πράσινο τουρισμό, για μικρές δηλαδή τουριστικές μονάδες, αλλά η πάση περιπτώσει να δαπανηθούν τα χρήματα αυτά με πολύ ξεκάθαρο τρόπο για έναν άλλο, ένα άλλο είδος ανάπτυξης. Και επανέρχομαι όχι μόνο στο θέμα του, το εμπορικό, αλλά δούμε και ένα τρίτο σημείο στα πλαίσια της πρότασης της Κομισιόν. Βλέπουμε πως ε, τα, οι επιπτώσεις γενικές, όπως ας πούμε επιπτώσεις στη διατήρηση του περιβάλλοντος, ε, με εντυπωσίασε ότι δεν είδα, μιλήσαμε μάλλον για την μπανάνα, αλλά δεν μιλήσαμε για το κλερντεκόν, δηλαδή για το... εκτός και αν αυτό δεν χρησιμοποιείται στην Καραϊβική. Με βάση αυτά που γνωρίζω είναι ότι οι μελέτες που αφορούν τις επιπτώσεις των φυτιών μπανάνας και ειδικά του, της χρήσης αυτού του κορντεκόν στις φυτίες μπανάνας αποτελεί κίνδυνο για την υγεία των ανθρώπων που εργάζονται στις φυτίες αλλά και μετά η γη δεν ήταν αρκετά καθαρή και κατάλληλη για άλλου είδους καλλιέργειες. Αν μιλάμε λοιπόν για αποκατάσταση του περιβάλλοντος και για διαφοροποίηση και για αλλαγή καλλιεργιών. Ε, νομίζω πως αυτό θα πρέπει να επιμείνουμε για να αποκατασταθεί όντως το περιβάλλον αλλά και να γίνει πραγματική ε, διαφοροποίηση στις καλλιέργειες. Μια τελευταία παρατήρηση. Διάβασα στη διαδικασία σε σχέση με τον τρόπο με τον οποίο θα εξεταστεί αυτό το θέμα, πρόκειται για συναπόφαση, Όλο ότι υπάρχει προαιρετική διαβούλευση με την Επιτροπή των Περιφερειών, πράγμα που για μένα σημαίνει τη σύνδεση με, με τα περιφερειακά συμβούλια. Ποια είναι η σύνδεση λοιπόν, αν υπάρχει, και πώς θα ληφθούν υπόψη όλα αυτά στη συνέχεια της ε, εξέτασης του θέματος. Σας ευχαριστώ. Ε, το λόγο έχει ο κύριος Μαρτίνες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Λίγα σχόλια Θέλω να ευχαριστήσω τον ε, ομιλητή γιατί μου φαίνεται, μου φαίνεται ότι μπόρεσε να διευκρινίσει πολλά σημεία σε αυτή την ε, υπόθεση και ο κύριος Γκέρανς επίσης. Καταρχήν, εγώ έρχομαι στο τελευταίο ερώτημα της κυρίας Γκρές. Θα ήθελα να ξέρω λοιπόν μέσα στο πλαίσιο που μας παρουσιάζονται, μας παρουσιάζει ο κύριος Μορασάν και η Κομισιόν, ποιος θα πρέπει να είναι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο εμπόριο ε, μπανάνας, συγκεκριμένα όμως για την ίδια παραγωγή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την παραγωγή σε υπερπεριφερειακές περιοχές, κάτι το οποίο σημαίνει Κανάρια, Μαδέρα, Ρεϊνιό, Μαρτινίκα, τα κτλ. Ποια είναι η διάσταση της ε, παραγωγής και της κατανάλωσης στο εμπόριο της μπανάνας που είναι ενδογενής, που παράγεται μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα λοιπόν η Κομισιόν να μας δώσουν μια επαλήθευση για τα μέτρα υποστήριξης που είναι πολύ σημαντικά για τις παραγωγές αυτές, για να μπορούμε να δούμε κατά πόσο μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την κινητοποίηση που γίνεται πολλές φορές σε αυτές τις περιοχές που θεωρούν ότι την χάνουν θύματα των ε, λεγόμενων ολεθρίων συμφωνιών στα πλαίσια του ΠΟΕ, ολέθριε σε σχέση με το μέλλον των περιοχών αυτών. Εγώ βέβαια δεν θέλω να υποστηρίξω μια τέτοια αντιμετώπιση θύματο από την πλευρά των παραγωγών στι περιοχέ αυτέ. Τώρα, για αυτά που είπε ο κ. Μορασάν σε σχέση με τι χώρε ΑΚΕ. Θα ήθελα να ξέρω αν έχει πραγματικά νόημα να μιλάμε για τι χώρε ΑΚΕ σαν να είναι μια ενιαία ομάδα χωρών. Γιατί σε ό,τι αφορά την μπανάνα, είναι φανερόν ότι είναι απόλυτα διαφοροποιημένη η κατάσταση των χωρών της Καραϊβικής έναντι των μεγάλων παραγωγών στην Αφρική, των οποίων η κατάσταση μοιάζει πολύ περισσότερο με τις μεγάλες χώρες παραγωγής στη Λατινική Αμερική και πολύ διαφορετική από αυτή των χωρών της Καραϊβικής. Ο κ. Μουρασάν είπε κάτι το οποίο μου φάνηκε πολύ σημαντικό. Είπε ότι στην Καραϊβική η παραγωγή μπαταμπανανών αφήνει ένα σημαντικά μεγαλύτερο ποσοστό προστιθέμενης αξίας στον παραγωγό και συγκεκριμένα σε αυτούς οι οποίοι εργάζονται στην καλλιέργεια και τη συγκομιδή. Είτε είναι ιδιοκτήτες είτε είναι εργαζόμενοι στον τομέα αυτό. Θα ήθελα όμως να έχω καλύτερα στοιχεία από την πλευρά του κυρίου Μόρασαν. Αναφέρθηκε ένα 11,5% σε γενικούς όρους πόσο είναι το ποσοστό αυτό σε άλλες περιοχές ΑΚΕ και συγκεκριμένα στην Καραϊβική και φυσικά πόσο είναι το ποσοστό αυτό στις μεγάλες τη περιοχή μεγάλη παραγωγή. Μια τελευταία παρατήρηση μου φαίνεται σημαντική επίση, κυρία Πρόεδρε, είναι η εξή. Εγώ τα τρία-τέσσερα χρόνια ή τα τελευταία δέκα χρόνια αρνήθηκα να υπησέλθω σε μια επιχειρηματολογία που διατυπώνεται από ορισμένου συναδέλφου και ιδίω από συναδέλφους που προέρχονται από πρώην απικιακές χώρες αυτοκρατορικού και υπεριαλιστικού χαρακτήρα χωρών κατά κάποιο τρόπο που ουσιαστικά φέρνουν αντιμέτωπα τα συμφέροντα των χωρών της Καραϊβικής με τα συμφέροντα άλλων χωρών πιο φτωχών, λιγότερο ανεπτυγμένες, που και λιγότερο ανεπτυγμένες από τις χώρες της Καραϊβικής. Νομίζω ότι εμείς θα πρέπει να είμαστε αλληλέγγυοι με το λαό της Καραϊβικής. Και θέλουμε πρώτα απ' όλα να υποστηρίξουμε την ανάπτυξη αυτής της περιοχής. Αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει δαιμονοποιώντας και καταδικάζοντας χώρες που βρίσκονται σε καταστάσεις οι οποίες είναι μεγαλύτερης ένδυας και μεγαλύτερης ανισότητος από ότι οι ίδιες οι χώρες της Δεν μπορούμε να πούμε ότι θα πρέπει να διατηρήσουμε αυτή την κατάσταση σε ορισμένες χώρες γιατί είναι χώρες που περιλαμβάνονται στη συνθήκη της Κοτονού αλλά δεν θέλουμε να γίνει αυτό να γίνει σε βάρος του να διατηρήσουμε σε πολύ μεγαλύτερη ένδια και αθλειότητα άλλες χώρες όπως χώρες της Κεντρικής Αμερικής που και αυτές έχουν ένα επίπεδο διαβίωσης το οποίο είναι πολύ υποδέστερο από τον χώρο της Καραϊβικής. Για μας η πρόκληση είναι να μπορέσουμε να εξισορροπήσουμε τη δράση μας με ένα τέτοιο τρόπο ώστε να επιτρέψει την ανάπτυξη και των μεν και των δε, δίνοντα την καλύτερη υποστήριξη στο εμπόριο τη μπανάνα, που είναι σημαντικό και για του με, για τους μεν αλλά και για του δε. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εμπειρογνώμονο μας, ε, κύριο Μορασάν και τον κύριο Γκέρενς για τι εξαιρετικά ενδιαφέρουσε ε, συμβολές τους. Να θέσω μια ερώτηση στον, κύριο, στον εμπειρογνώμονά μας όσον αφορά την κατανομή των ε, χρηματοπιστωτικών ροών ανάμεσα στους παραγωγούς, ε, τους διανομής και τις εταιρείες. Ε, λέγατε στην, εισήγηση, εισαγωγή σας ότι 40% χονδρικά πάει για τα σούπερ μάρκετ και το 36% για τις εταιρείες. Μπορέσατε να κάνετε διάκριση ανάμεσα στα κέρδη των εταιριών στις χώρες onshore και στις χώρες offshore. Μπορέσατε να δείτε πού δηλαδή πάνε τα... πού γίνονται μάλλον τα κέρδη της Τσικίτα και των άλλων. Συνολικά τρία ερωτήματα έχω να αντιμετωπίσω. Για την εγχώρια παραγωγή μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση η ανάλυση μου επικεντρώθηκε στο θέμα του εξωτερικού εμπόριου. Γι' αυτό δεν ασχολήθηκα με την εσωτερική παραγωγή τη Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί μιλούσαν περισσότερο για εισαγωγέ και εξαγωγέ. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν μελέτε σε σχέση με τι ενδεχόμενε επιπτώσει που θα μπορούσαν να προκύψουν από τη μείωση των δασμών που προφανώς προστατεύουν την εγχώρια παραγωγή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίση υπάρχουν μελέτες σε σχέση με την επίπτωση των συμφωνιών αναπτυξιακού και εταιρικού χαρακτήρα στην εγχώρια παραγωγή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό το οποίο έχει προκύψει είναι ότι ο αντίκτυπος της φιλελευθεροποίησης της, του καθεστώτος εισαγωγής για την εγχώρια παραγωγή στη Μαδέρα, στα Κανάρια, στην Κρήτη είχε, έχει ήδη λάβει χώρα. Δηλαδή αυτή η φιλελευθερωποίηση έλαβε χώρα με την ε, σταδιακή μείωση των δασμών. Αν υπάρξει λοιπόν περαιτέρω φιλελευθερωποίηση θα υπάρξει μια μικρή μονάχα ε, επίπτωση γιατί η πραγματική αλλαγή ήταν η κατάργηση των ποσοστώσεων από την 1η Ιανουαρίου 2007. Δεν βλέπουν λοιπόν οι εμπειρογνώμονες ότι αυτές οι συμφωνίες της Γενέβη θα έχουν σημαντικά αρνητική αντί... Ε, επίπτωση για την παραγωγή την εγχώρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα τώρα με αυτό που λέει ο κύριος Ματίνες, ήταν ένα τμήμα αυτών των πραγμάτων που ήθελα να πω, ότι είναι απαραίτητο να κάνουμε μια διαφοροποίηση αρκετά σαφή μεταξύ των ίδιων των χωρών που είναι στην ομάδα των χωρών ΑΚΕ. Η διαφοροποίηση αυτή έχει εδρεωθεί ήδη στην αγορά, στην Αφρική. Η Αφρική έχει δύο μεγάλους παραγωγούς ή μεγάλους εξαγωγείς και μία μεσαία χώρα είναι το Καμερούν και η ακτή του Αλεφαντοστού που είναι οι κύριοι κερδισμένοι της προστασίας της αγοράς τα τελευταία χρόνια και ενδεχομένως και η Γκάνα είναι και αυτή μια δυναμική αγορά η οποία αναδύεται αυτή τη στιγμή. Αλλά για την Καραϊβική. Και η Δομινικανική Δημοκρατία είναι τμήμα της Καραϊβικής και είναι ο πρώτος κερδισμένος από όλα αυτά τα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί την τελευταία αυτή δεκαετία. Ώστε η δημοκρατία, η δομινικανική, έχει αυτή τη στιγμή το 55% των εξαγών της σύνολης περιοχής της ε, Καραϊβικής. Επίσης ευνοήθηκε η Μπελίζε και το Σουρινάμ, όπως είπα, βάσει των εκτιμήσεων των εμπειρογνωμόνων, οι χώρες αυτές μάλλον θα μπορέσουν να αντέξουν το σοκ της φιλελευθερωποίησης παρά το γεγονό ότι χρειάζονται μια υποστήριξη για να βελτιώσουν ορισμένε ε, συνθήκες ό,τι αφορά την παραγωγή τη μπανάνα. να βελτιώσουν τι διεργασίε παραγωγή. χρειάζονται την υποστήριξη για να έχουν καλύτερη οργάνωση τη αγορά και καλύτερο μάρκετινγκ επίση. Αυτοί που θα χάσουν μέχρι στιγμή, οι μεγάλοι χαμένοι, είναι τα μικρά νησάκια, τα προσύνεμα νησιά, τα Windward Islands. Αλλά παρόλα αυτά μπόρεσαν να βρουν μια ειδική γονίτσα της αγοράς που είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε μια καλύτερη ανάλυση της ε, αλυσίδας αγοράς. Το 80% των εξαγωγών των χωρών αυτών είναι οι μπανάνες fair trade. Και νομίζω ότι έχουν επιτύχει ιδιαίτερα στον τομέα αυτό. Ήταν πολύ επιτυχής αυτή η διαδικασία και γι' αυτό θα ήταν απαραίτητο να γίνει μια μελέτη για τα μέτρα αυτά, όχι μονάχα της ε, εμποριοποίησης, αλλά και του πώς μπορεί κανείς να ευνοήσει και να αναβαθμίσει την αλυσίδα προσθέμενης αξίας της χώρες αυτές. Σε ό,τι αφορά την διαφορά που μου ζητήσατε να κάνω, να διαφοροποιήσω, νομίζω ότι όπως είπε και ο κ. Μαρτίνες υπάρχει μια σημαντική διαφορά σε ό,τι αφορά έσοδα και ημερομίσθια μεταξύ κάποιου που εργάζεται στον Ισημερινό και ε, κάποιου που δουλεύει στο Καμερούν. Αλλά Υπάρχουν μεν, αλλά είναι πολύ μικρές αυτές οι διαφορές. Το πρόβλημα το οποίο τίθεται είναι ότι από τη δεκαετία του 1990 υπάρχει μια αλλαγή σε ό,τι αφορά την ισχύ που έχουν οι διάφοροι παίκτες στην αλυσίδα προσθέμενης αξίας, ακόμα και στην περίπτωση που αυτή είναι ενσωματωμένη και ολοκληρωμένη και ο κερδισμένος αυτή τη στιγμή είναι τα σούπερ μάρκετ που καθορίζουν τις τιμές και αποκομίζουν τη μερίδα του λέοντος στο, στα κέρδη αυτά, είτε πρόκειται για τη ζώνη του δολαρίου ή για τη ζώνη των χωρών και αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα το οποίο αξίζει να το εξετάσουμε γιατί εάν εμείς θεωρούμε, πολλοί εμπειρογνώμονες το θεωρούν, ότι πράγματι είναι δυνατόν μέσα από μέτρα συνοδευτικού χαρακτήρα να επιτύχουμε να γίνουν οι απαραίτητες <clears throat> αλλαγές στην πολιτική μας ανάπτυξη ώστε η έλλειψη ισορροπίας στην αλυσίδα προσθέμενης αξίας σε βάρος των παραγωγών να αντισταθμιστεί από μέτρα τα οποία είναι ε, συμβατά με την αγορά, συγκεκριμένες παρεμβάσεις λοιπόν που δεν έχουν προστατευτικού χαρακτήρα, αυτό πιστεύουμε ότι τότε πρέπει να γίνει. Ευχαριστώ πολύ. Κύριος Βέγγελ. Σα Σας ευχαριστώ. Είναι ξεκάθαρο για μένα γιατί μιλάμε για την παραγωγή μπανάνας και το εμπόριο μπανάνας σε τέτοιο βαθμό και συμφωνώ πως είναι πολύ ενδιαφέρουσα και σημαντική η συζήτηση για ένα σωρό χώρες. Αυτό όμως το οποίο λείπει από τη συζήτηση είναι ένα συστατικό που νομίζω πως επίσης έχει τη σημασία του. Σε ολόκληρη την αλυσίδα τροφίμων και αν δει κανεί ε, την κατανάλωση τροφίμων σε ολόκληρο τον κόσμο, θα πρέπει να δούμε τι έχουν σημάνει τα τελευταία 10 χρόνια για με την παραγωγή μπανάνας. Φαντάζομαι πως αυτό δημιουργεί κάποια προστιθέμενη αξία για ορισμένους, αλλά αφαιρεί προστιθέμενη αξία από κάποιους άλλους. Οι ευκαιρίες ε, για ε, προστιθέμενη αξία στο πλαίσιο της βιοπικιλότητας επίσης. Ιδιαίτερα όσον αφορά τη διατροφική διαφοροποίηση. Και θα ήταν ενδιαφέρον, οποτεδήποτε συζητούμε πολιτικές στήριξης, για χώρες τις οποίες στηρίζουμε με τον τρόπο αυτό και μέσω της εργασίας της δικής μας Επιτροπής, θα ήταν καλό να συμπεριλαμβάνουμε ένα επιπλέον στοιχείο στη συζήτηση αυτή για το τι δηλαδή ακριβώς σημαίνει η παραγωγή μπανάνας όσον αφορά την διατροφική της αξία. Και να σας πω, να σκεφτούμε μάλλον επίσης ότι η υπερβολική δίκευση στην καλλιέργεια μπανάνας αποκλείει αυτές τις χώρες από το να έχουν καλύτερα αποτελέσματα με άλλα προϊόντα, φρούτα ή άλλα γεωργικά προϊόντα εν γέννη. Ίσως αυτή η ιδέα να μην είναι και στο επίκεντρο του σημερινού θέματος, αλλά σίγουρα δεν είναι και τελείως άσχετη. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει τώρα η Κομισιόν, που την οποία αντιπροσωπεύει ο κύριος Λουί Γκριγέρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομος, γιατί νομίζω πως υπάρχουν πολλά, τα οποία ήδη υπόθηκαν. Να σας ευχαριστήσω καταρχήν που μας δίνετε την ευκαιρία να πάρουμε το λόγο και να ευχαριστήσω τον κύριο Γκέρενς που διοργάνωσε αυτή τη συζήτηση και που ζήτησε να γίνει αυτή η μελέτη, η οποία πραγματικά φωτίζει ένα εξαιρετικά περίπλοκο θέμα, μια εξαιρετικά περίπλοκη αγορά. Να ευχαριστήσω και τον εμπειρογνώμονά μας. Ελπίζω πως θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε κάποια από τα πορίσματά σας αργότερα. Νομίζω πως συμφωνούμε πλήρως όσον αφορά, τόσο όσον αφορά τη διάγνωση όσο και τις προτάσεις, τις λύσεις. Συμμεριζόμαστε την άποψη πως η κατάσταση είναι εξαιρετικά διαφορετική στις χώρες ΑΚΕ, ανάμεσα στις διάφορες χώρες ΑΚΕ και γι' αυτό και θα πρέπει να δοθούν διαφοροποιημένες απαντήσεις. Και όταν κανείς εξετάσει τα τρία είδη δράσεις που έχουμε προτείνει, Νομίζω πως αυτά συμπίπτουν ακριβώς με το είδος των συστάσεων που έχετε προτείνει. Είναι αλήθεια, όπως είπε και ο κύριος Μαρτίνες, πως πρόκειται για εξαιρετικά περίπλοκο τομέα όπου κατά κάποιο τρόπο πρέπει να συνδυάσουμε πολλά διαφορετικά συμφέροντα. Ειλικρινά πιστεύω πως έχουμε μια καλή ισορροπία με τη Συμφωνία της Γενέβης. Οι χώρες ΑΚΕ γνώριζαν ότι θα γινόταν αυτή η κατάργηση των εμπορικών φραγμών. Αλήθεια είναι ότι ίσως έγιναν πιο σύντομα από ό,τι περίμεναν όλα αυτά. Και γι' αυτό και πιστεύουμε πως πρέπει να βοηθήσουμε περαιτέρω την προσαρμογή των χωρών αυτών. Και νομίζω πως αυτά που κάναμε με βάση τα προηγούμενα προγράμματα έδωσαν, προσέφεραν μια καλή βάση για να βοηθήσουμε τις ε, χώρες αυτές. Είναι αλήθεια, όπως υπόθηκε, ότι θα πρέπει να ότι μαθαίνουμε από την εμπειρία μας Όντως, τα μέτρα διαφοροποίησης που χρησιμοποιήθηκαν στο παρελθόν δεν έδωσαν πάντοτε τα αποτελέσματα που περιμέναμε. Ούτε εμεί τα κρατημέλη, ούτε και οι χώρες δικαιούχοι όλων αυτών των προγραμμάτων. Ίσως γιατί όντως δεν στοχεύσαμε την στήριξή μας ε, επαρκώς. Και ένα από τα βασικά μενήματα που έχουμε αποκομίσει από τη μελέτη που έχουμε κάνει και για να αναλύσουμε κάπως ε, το βασικό αντίκτυπο της παλαιότερης ενίσχυσης είναι ότι όντως θα πρέπει να είμαστε πολύ πιο στοχευμένοι στο μέλλον και ιδιαίτερα για τις χώρες που βρίσκονται στη μέση και που μπορεί με κάποια στήριξη να διατηρήσουν μια ανταγωνιστικότητα στο ευρωπαϊκή αγορά, αλλά χρειάζονται κάποια διαφοροποίηση. Και είναι αλήθεια πως τα μέτρα διαφοροποίησης πιθανότατα δεν ήταν αρκετά καλά ε, αρκετά μάλλον στοχευμένα και αυτό μας ε, δίνει καλή εμπειρία για το μέλλον. Ο εμπειρογνώμονες μίλησε για αντίκτυπο στις ευρωπαϊκές χώρες. Ε, με τις αναλύσεις που έχουμε κάνει πιστεύουμε πως η ο βασικός αντίκτυπος έχει ήδη περάσει και με μια μεγάλη αύξηση στην ε, κατανομή των θέσεων μπορούμε να διασφαλίσουμε την ανταγωνιστικότητα των εγχώριων παραγωγών μας. Λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη το θέμα όσον αφορά το περιβάλλον και νομίζω πως ε, αυτό θα πρέπει να προσεχθεί πολύ ιδιαίτερα για τις χώρες που μπορεί να ακολουθήσουν τον δρόμο της διαφοροποίησης κάποιου τμήματος της παραγωγής τους. Αυτά είχα να πω σε αυτό το στάδιο. Ίσως μία ακόμα παρατήρηση στον συνάδελφο που έκανε τη μελέτη δεν, μπορούμε, δεν, δεν θέλουμε να φτάσουμε στην μηδενικό δασμό, ε, όπως γνωρίζετε, για τις χώρες οι οποίες τώρα έχουν ε, ε δασμό MFN. Θα φτάσουν στο 114% το 2017. Για τις χώρες από την Λατινική Αμερική που μπαίνουν ε, στην, ε, τρίτη, στη φάση fair trade θα φτάσουν σε, χαμηλότερο δασμό μέχρι το 2020, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα υπάρχει μηδενικός δασμός. Νομίζω ειλικρινά πως έχουμε φτάσει σε μια καλή ισορροπία σε μια τόσο περίπλοκη κατάσταση και προσβλέπουμε συνεργασία μαζί σας και με, ειδικά με τον κύριο Γκέρενς γιατί όπως είπαμε είναι ένα συνολικό πακέτο και θα προσπαθήσουμε να προχωρήσουμε με παράλληλα σε όλα τα μέτωπα, γιατί διαφορετικά κινδυνεύουμε να θέσουμε σε κίνδυνο ολόκληρο το πακέτο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κι εγώ. Κύριε Γκέρενς, έχουμε αργήσει πάρα πολύ. Κυρία Γκρικεζέρ που πρέπει να φύγει σύντομα, που έχει το επόμενο σημείο. Γι' αυτό σας παρακαλώ να είστε πολύ σύντομος στα συμπεράσματά σας. Σας ευχαριστώ. Να πω δύο λόγια απαντώντας σε όσους ε, παρενέβηκαν. Στην κυρία Γκρέας να της δώσω δύο απαντήσεις. Η πρώτη αφορά τα ζενοκτώνα, το κλόρντεκόν. Εκεί θα πρέπει να εφαρμοστεί η αρχή του ρηπαίνων πληρώνει. Ε, δηλαδή δεν είναι θέμα το οποίο θα πρέπει να επιβαρύνει το κοινοτικό προϋπολογισμό. Εφόσον πρέπει να γίνει αποκατάσταση γεών, αυτό θα πρέπει να επιβαρύνει τους ε, ρηπαίνοντες. Το κονδύλι το οποίο θα δοθεί θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για να γίνει διαφοροποίηση των καλλιεργειών. Εδώ βλέπω δύο οδούς. Διαφοροποίηση σημαίνει και μεταποίηση της μπανάνας επιτόπου. Μπορούν να γίνουν πολλά προϊόντα με βάση αυτή την πρώτη γιατί αυτό να μην γίνει επιτόπου παρά να γίνεται στις χώρες ε, κατανάλωσης και έπειτα. Αν αυτή η διαφοροποίηση είναι δύσκολο να γίνει, να υλοποιηθεί, θα μπορούσαμε να δούμε μια, μια αλλαγή κατεύθυνσης παραγωγής προς άλλους τομείς. Νομίζω πως ε, αυτά τα κονδύλια λοιπόν θα μπορούσαν να δοθούν στη μία ή στις δύο κατευθύνσεις ή και στις δύο ταυτόχρονα. Δεύτερον, αναφέρατε τα υπερπόντια εδάφη. Η κατάσταση φυσικά έχει αλλάξει στο βαθμό που η μία και πιο εύκολα θα φτάσουν στις αγορές μας. Θα θυγούν ωστόσο και, όπως και η ΑΚΕ. Θα πρέπει να δούμε και να κινητοποιήσουμε άλλα κονδύλια για να αντιμετωπιστούν τα δικά τους προβλήματα. Και έπειτα, κύριε Μαρτίνες, να μην ζημιωθούν τα συμφέροντα των όσων δεν έχουν ε, προστάτευες δυνάμεις, αν κατάλαβα καλά το μήνυμά σας. Υπάρχουν τρεις κατηγορίες ε, εξαγωγικών ε, χωρών μπανάνες. Στη μία και η ΑΚΕ και εντός των ΑΚΕ υπάρχουν ε, η Καραϊβική και η Νότια Αφρική. Η μία ΑΚΕ έχει βελτιωθεί η κατάστασή τους. Ανάμεσα στους ΑΚΕ οι λατινοαμερικανικές χώρες διατηρούν μεγάλο πλεονέκτημα έναντι της Αφρικής γιατί έχουν μια αγορά στη, <laughs> στα σύνορά τους πολύ πιο προσβάσιμη Υπάρχει ένα θέμα μεγέθους, το οποίο δεν ανέφερα, είναι η δυσκολία των Αφρικανών να μπουν στην, να διεισδύσουν στην Αμερικανική αγορά. Ε, α, απουσιάζουν από τις Αμερικάνικες αγορές. Και τελευταία παρατήρηση, και το διαπίστωσα και στις συνομιλίες που είχαμε την Κομισιόν, ότι η Κομισιόν είναι ένα μέρος του προβλήματος, αλλά είναι και μέρος της λύσης, γιατί εδώ αμφισβητείται το καθεστώς ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης εδώ και 15 χρόνια, για πόσους δικαίους ή αδίκους θεωρούν ότι δικαίως ή αδίκως θεωρούν ότι ζημιώνονται από τις προτιμησιακές πρακτικές που, ε, που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση με ορισμένες χώρες. Κρίμα που δεν έχουμε αρκετό χρόνο, αλλά είμαι έτοιμος να θυσιαστώ για την κυρία Ντικεζέρ. Euh, euh, και τώρα θα περάσουμε στο επόμενο σύστημα της μέσης διάταξης, τα συστήματα υγείας στην υποσαχάρια Αφρική. Έχουμε αποφασίσει να κάνουμε μια έκθεση πρωτοβουλία για αυτό το σημαντικό θέμα και δίνω το λόγο στην κυρία Ντεκέιζερ Οσονούπο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον κύριο Γκέρετς για την αυτοθυσία του. Εγώ πρέπει να θυσιαστώ για τη Βελική Προεδρία γιατί λαμβάνει η χώρα στο Παλέντεγμό μια συνεδρία που αρχίζει σε ένα τέταρτο είχαμε κάνει μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων για αυτή την έκθεση, την οποία εγώ θα ήθελα τώρα να παρουσιάσω σε εσά, μάλλον η πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Αυτό το οποίο θα σας παρουσιάσω εντάχει είναι η στόχη αυτής της έκθεσης που σε μεγάλο βαθμό έχει ήδη συγγραφεί, αλλά θα ήθελα να έχω και τις απόψεις σας για να την κατευθύνω με το σωστό τρόπο. Καταρχήν έχουμε μία διαπίστωση η οποία είναι τρομακτικού χαρακτήρα, ότι δηλαδή Υπάρχει ένα πραγματικό χάσμα που χωρίζει τους Ευρωπαίους από τις υποσαχάριες αφρικανικές χώρες. Η διαφορά σε προσδόκιμο επιβίωσης μπορεί να είναι 30-40 χρόνια κιόλα. και υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες οι οποίοι μπορούν να αιτιολογήσουν αυτή τη διαφορά. Φυσικά υπάρχουν οι μεγάλες επιδημίες, η ελονοσία, το AIDS κτλ. Αλλά κυρίως και η ένδια, <clears throat> η υπανάπτυξη της Αφρικανικής Υπήρου, η κακοδιακυβέρνηση πολλών χωρών, τα αποτελέσματα της χρηματοοικονομικής κρίσης που οδήγησαν σε μεγαλύτερη επιδείνωση της ένδυας στις χώρες αυτές και η κλιματική αλλαγή, άμα τα βάλουμε όλα αυτά μαζί, καταλήγουμε σε μια τρομακτική διαπίστωση. Η Επιτροπή μας έχει τονίσει το πόσο σημαντικό να υπάρχουν αυτά τα κάθετα ταμεία τα οποία μπορούν να βοηθήσουν τις χώρες αυτές. Ξέρουμε όμως είναι και ποια είναι τα όρια τους. Δίνουν αποτελέσματα τα οποία είναι αδιαμφισβήτητα, αλλά συγχρόνως θα πρέπει εμείς στην Αφρική να δημιουργήσουμε τις λεγόμενες οριζόντιες μορφές υγειονομικής περίθαλψης, όχι μοναχα κάθετες, γιατί είναι γεγονός ότι οι κύριες αιτίες θανάτου Μπορεί να είναι οι μεγάλες επιδημίες, αλλά υπάρχει και ένα υπόβαθρο θνησιμότητος που οφείλεται σε προβλήματα περίθαλψης, σε περίπτωση εγκυμοσύνης, δύσκολης κοίησης, για ασθένειες που δεν μπορούν να θεωρηθούν ότι είναι καθημερινές ασθένειες, αλλά είναι ασθένειες που προκύπτουν από την ένδυα και την αθλειότητα. Επομένως, η ιδέα που διατρέχει αυτή την έκθεση είναι ότι αυτές οι οριζόντιες παροχές υγειονομικής περίθαλψης θα πρέπει να ενισχυθούν και να χρησιμοποιηθεί η διεθνής βοήθεια προς το σκοπό αυτό. Όταν εξετάζουμε τώρα τη χρηματοδότηση αυτών των οριζοντίων μορφών περίθαλψης, βλέπουμε ότι τα, οι κάθετες μορφές περίθαλψης καταλαμβάνουν ένα μεγάλο μερίδιο της παγκόσμιας βοήθειας και της προσοχής των φιλανθρωπικών οργανώσεων, ενώ στην περίπτωση τη οριζόντιας περίθαλψης είναι πολλά τα οποία παραμένουν να γίνουν και δεν μπορούμε να φανταστούμε ότι σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα μπορούν αυτέ οι υπηρεσίε να έχουν ένα βιώσιμο χαρακτήρα μόνο με τι προσπάθειε των κρατικών προπολογισμών. Γι' αυτό λοιπόν και αυτή είναι η ουσία τη έκθεση, γι' αυτό είναι σημαντικό να επικεντρώσουμε την προσοχή μα προ μια χρηματοδότηση η οποία θα ερχόταν από τους ίδιους τους πληθυσμούς εγώ έδωσα μεγάλη σημασία στις πρωτοβουλίες οι οποίες ξεκίνησαν τη δεκαετία του 90 στην Αφρική για όλα αυτά τα συστήματα ε, ασφαλιών, μικροασφαλίσεων. Αυτά τα συστήματα λοιπόν τα οποία έχουν πολλαπλασιαστεί με τρόπο ο οποίος είναι κάπως λίγο άναρχος ακόμα και όχι ιδιαίτερα συντονισμένος αλλά που βασίζονται σε μια βασική ακόμα αξία στην Αφρική που είναι η αρχή της αλληλεγγύης και της αλληλοβοήθειας. Ξέρετε ότι υπάρχει αυτός ο μηχανισμός στην Αφρική όταν κάποιος σε ένα χωριό ή σε μια φίλη έχει ένα πρόβλημα υγείας, όλοι δίνουν υπομορφή ρεφενέ για να μπορέσουν να τον βοηθήσουν να πάει στο γιατρό στο νοσοκομείο. Αυτό ισχύει σε όλες τις ε, φυλές της Αφρικής. Επομένως θα μπορούσαμε να το χρησιμοποιήσουμε αυτό όχι για να γίνεται αυτή η συλλογή χρημάτων, αυτό το είδος εράνου, για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα κάποιου, αλλά για να υπάρχουν κάποια ποσά τα οποία θα μπορέσουν να καλύψουν μια μορφή προληπτική ιατρική. Να μπορούμε λοιπόν σιγά σιγά να προβλέψουμε να δημιουργηθεί ένα σύστημα υγειονομική ασφάλισης το οποίο να είναι βιώσιμο. Αυτό το οποίο είναι πολύ σημαντικό και ενδιαφέρον είναι ότι σε πολλέ χώρε τη Αφρική έχουν ξεκινήσει τέτοιου ε, εμπειρίε και πειράματα η, τα δημοκρατική, η δημοκρατία του Κονγκό, Μπουρκίνα Φάσο, Μπουρούντι, Κονγκό, ε, Σενεγάλη μάλλον, το πράσινο ακροτήριο και με τη βοήθεια πολλές φορές των μη κυβερνητικών οργανώσεων αλλά και με ευρωπαϊκούς ασφαλιστικούς φορείς που έχουν παραδείγματος χάρη χριστιανικό χαρακτήρα ή σοσιαλιστικό χαρακτήρα και έχουν προσπαθήσει σε τοπικό επίπεδο ή σε εθνικό επίπεδο, ακόμα και σε διεθνές επίπεδο, να οργανώσουν καλύτερα το σύστημα αυτό <clears throat> της αλληλοβοήθειας, ώστε να καταλήξουμε σε μία μορφή εναλλακτική χρηματοδότησης η οποία μπορεί να υποστηρίξει τα συστήματα αυτά τα οποία αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να σταθούν πολύ καλά στα πόδια τους. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά σε κοινωνικό επίπεδο γιατί βασίζονται σε αρχές ενδογενή στην Αφρική και μας δίνει και μας την έννοια της αλληλεγγύης βορρά-νότου με μια διαφορετική μορφή. Αυτές λοιπόν είναι οι βασικές ιδέες που περιέχονται στην έκθεσή μου, που εστιάζουν την προσοχή τους στις μορφές αυτές αλληλοβοήθειας και περιέχει επίσης η έκθεση μια σειρά από συστάσεις προς την Κομισιόν σε ό,τι αφορά τα οριζόντια συστήματα υγείας, γιατί πρέπει να σκεφτείτε <clears throat> ότι οι πληθυσμοί ήδη φυσικά έχουν κάποια χρήματα τα οποία χρησιμοποιούν για να βοηθήσουν τους ε, ασθενείς και τους αρρώστους. Δεν θα το κάνουν αυτό όμως παρά μόνο αν υπάρχουν φάρμακα και νοσοκομεία στην περιοχή τους ώστε να μπορούν να έχουν αυτή την περίθαλψη. Φυσικά θα πληρώσουν εάν δεν υπάρχουν οι υποδομές για να του περιθάλψουν. Λοιπόν, αυτή η δυναμική μεταξύ των συστημάτων οριζόντια περίθαλψη και τη ανάπτυξη αυτή τη μορφή αλληλοβοήθεια και ε, είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον γιατί αυτό μα επιτρέπει να δούμε στο μέλλον να αναδύεται κάτι το πιο βιώσιμο το οποίο βασίζεται στι τόσο σημαντικές αρχές αλληλεγγύη, σημαντικέ για την Αφρική και αυτό θα μπορούσε να είναι ένα υπόδειγμα το οποίο θα συμπληρώνει τις ε, προσπάθειες που γίνεται πολλές φορές σε επίπεδο επίγουσας ανακούφισης από τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις, γιατί η Αφρικανική Ήπειρος μαστίζεται από τις συγκρούσεις, υπάρχουν μη κυβερνητικέ οργανώσεις που δίνουν δωρεάν περίθαψης βοηθούν τους πληθυσμούς, αλλά ξέρουμε ότι αυτή η μορφή κατεπίγουσας βοήθειας και αυτή η μορφή δωρεάν βοήθειας δεν είναι αυτό το οποίο θέλουμε να αναπτυχθεί, διότι θέλουμε να δώσουμε την δυνατότητα στην Αφρική να αναπτυχθεί με έναν τρόπο ο οποίος είναι ισότιμος και αυτόνομος εν καιρό και επομένως και εν καιρό βιώσιμος. Αυτές λοιπόν είναι οι βασικές κατευθυντήριες γραμμές της έκθεσής μου, του πρώτου σχεδίου της έκθεσής μου. Ήλπιζα να την έχω μεταφρασμένη εδώ σήμερα, αλλά δεν είναι γεγονός αυτό αλλά είμαι έτοιμη μαζί με την ομάδα μου, μαζί με τη γραμματεία μου, να ακούσω τις απόψεις σας, τα παραδείγματα που θέλετε να μου δώσετε, την κάθε μορφή υποστήριξης, αλλά ήθελα προς να σας εξηγήσω ποια ήταν η δική μου οπτική γωνία, η εναρκτήριά μου προσέγγιση και η οποία πιστεύω ότι μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο συνένεση μεταξύ των πολιτικών ομάδων. Αυτά λοιπόν θέλω να πω κυρία Πρόεδρε και σας ευχαριστώ και θα ακούσω με μεγάλη προσοχή αυτά που έχουν να πούν οι συναδελφοί μου. Ο κύριο Μίντζελ έχει ζητήσει το λόγο. Κυρία Πρόεδρε, θα είμαι πολύ σύντομο. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Τεκεζέρε για την έκθεσή τη. Δεν έχω αντίγραφό τη, ίσω να το έχω στο γραφείο μου, αλλά εγώ δεν την έχω την έκθεση μπροστά μου. Ελπίζω πως να υπάρχει γενικά συνένεση στα θέματα που προκύπτουν από αυτή την έκθεση. Όλοι ανησυχούμε για την ελονοσία, το AIDS και ανησυχούμε ε, και θα έπρεπε, όπως θα έπρεπε εξάλλου και θα, είναι θέματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Να πω μόνο πως ε, σοκαρίστηκα πριν από λίγες εβδομάδες γιατί παρακολούθησα μία παρουσίαση για τις μη μεταδοτικές ασθένειες στον απτυσσόμενο κόσμο και να δω, εδώ ανακαλύψω για παράδειγμα ότι τα καρδιακά επεισόδια σε σχέση με πίεση ή εμφράγματα, δηλαδή ασθένειες στις οποίες είμαστε συνηθισμένοι στη Δύση δεν είναι πολύ πέρα στη κλίμακα Ρίχτερ. Δεν συμβάλλουν, ε, δεν, δεν έχουν σημασία. Ε, δεν τα εξετάζουμε αυτά τα νοσήματα όπως ε, τις μεταδοτικές ασθένειες. Πρέπει δηλαδή να εξετάσουμε ποιο είναι το αίτιο, ποιο είναι το αίτιο θανάτου ασθένειας ή πόνου, ό,τι και αν είναι αυτό, και να προσπαθήσουμε να βρούμε μια λύση με τον τρόπο με τον οποίο παρουσίασε η κυρία Ντεκάζη. Δεν γνωρίζω ακόμα το πλήρες περιεχόμενο της έκθεσης, αλλά σίγουρα πρέπει να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να δώσουμε σωστές υπηρεσίες υγείας στον αναπτυσσόμενο κόσμο. Αν θυμάμαι καλά, ιδιαίτερα τα καρδιακά επεισόδια στις γυναίκες ήταν τεράστια. Ε, το ποσοστό. Δηλαδή ήταν εδώ κάτω το AIDS και η ελονοσία, ενώ τα καρδιακά επεισόδια ήταν εκεί πάνω. Πρέπει να δούμε λοιπόν την έκθεση και να ελπίζω να μπορέσουμε να φτάσουμε σε συνένεση για το περιεχόμενο. Να προσπαθήσουμε να δώσουμε στον κόσμο που το χρειάζεται πραγματικά πρόληψη και θεραπεία. Όπως αυτές που έχουμε εδώ στον αναπτυγμένο κόσμο. Ευχαριστώ, κύριε Γκέρενς. Ευχαριστώ. Δεν θα φάω το χρόνο, ελπίζω, της κυρίας Τεκέιζερ. Έχουμε λοιπόν τους στόχους για την ανάπτυξη και διαπιστώνουμε σε πάρα πολλές χώρες δεν υπάρχει ε, σαφής φιλοδοξία για να ε, εξασφαλιστούν ε, οι διατάξεις και τα κονδύλια για να μπορέσει κανείς να πετύχει αυτούς τους στόχους. Λοιπόν, ήθελα να πω το εξή. Αυτό που είναι σημαντικό είναι να έχουμε από τη μια έχουμε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν τίποτα, δεν μπορούν δηλαδή να χρηματοδοτήσουν συστήματα ασφάλειας για να καλύψουν τα, τις δαπάνες για ένα σύστημα για την προστασία της υγείας. Έχουμε το συνολικό, τα συνολικά κονδύλια που αφορούν το καταπαλισμό της φυματίωσης, της ελονοσίας και άλλων ασθενειών. Αυτό που είναι σημαντικό, οι χώρες αυτές να εντάξουν τους προβληματισμούς που αναφέρει η κυρία Ντεγκέιζερ για, το, για τη μελλοντική τους ανάπτυξη. Έχουμε λοιπόν την εσωτερική εταιρική συνεργασία. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την, ε, την συμβολή εμπειρογνωμόνων και φυσικά προσπάθειες τόσο σε επίπεδο ε, Ηνωμένων Εθνών και άλλων διεθνών συνεργασιών να προχωρήσουμε. Επίσης να δούμε και τη διάσταση που έχει να κάνει σε περιφερειακό επίπεδο. Βλέπουμε τη, τον Ήγηρα. Σε, σε απόσταση φέρει πέν. Έχουμε για παράδειγμα, βλέπουμε ας πούμε, στην Ελλάδα του Νίγηρα, ότι 30 χιλιόμετρα πιο δυτικά τη σημεία όχθη υπάρχει μια δραστηριότητα και το ίδιο από την άλλη απόσταση, χωρί να υπάρχει μια οποιαδήποτε συνεργασία. Ε, θα πρέπει λοιπόν να δούμε ποιες είναι οι ανάγκες επιτόπου και να προβλέψει κανείς τις κατάλληλες υποδομές. Επίσης, εν ώψη των διαπραγματεύσεων για το διεθνές εμπόριο σεβόμενοι και τις διατάξεις που σύρουν για την εργασία σε διεθνές επίπεδο να κοιτάξουμε να προωθήσουμε το εμπόριο των χωρών της Αφρικής και να σκεφτούμε ότι οι χώρες της Αφρικής που έχουν λίγες, μικρή απόδοση όσον αφορά την εμπορική ανάπτυξη πτήξη για να μπορέσουν να πετύχουν Φερπίν μια εξαγωγική πολιτική χρειάζεται να βοηθηθούν οι παραγωγοί, θα πρέπει να γίνονται επενδύσεις ε, σε νέα προϊόντα και φυσικά σημαίνει αυτό ότι θα πρέπει να πάρει κανείς και ένα ρίσκο. Ε, και αυτό το ρίσκο έχει τις επιπτώσεις όσον αφορά και την κοινωνική ασφάλεια. Και έτσι δημιουργείται ένας ε, φαύλος κύκλος. Όταν δεν έχεις το ένα δεν έχεις το άλλο και τα ανάπαλη είναι. Χρειάζεται δηλαδή από τη μια ε, η ανάπτυξη μπορεί να οδηγεί σε κοινωνική προστασία, αλλά από την άλλη χρειάζεται κοινωνική προστασία για να μπορέσει κανεί να επενδύσει και να εξασφαλίσει καλύτερε συνθήκε για την εμπορική του ανάπτυξη. Ευχαριστώ, Πρόεδρο. Ευχαριστώ. Ο κύριο Καρέ, εκ μέρου τη Επιτροπή, θα πάρει το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Εμείς δεν έχουμε καταφέρει ακόμα να δούμε το σχέδιο έκθεσης και προσβλέπουμε στο να το δούμε. Η πρώτη μου αντίδραση θα ήταν ότι ελπίζω ότι η συγγήτρια έχει λάβει υπόψη την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα θέματα υγείας, είναι ένα έγγραφο το οποίο διαβάστηκε στο Κοινοβούλιο και φυσικά και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου στις 10 ε, Μαΐου για το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υγεία στην Ήπεθρο. Νομίζω ότι είναι σημαντικό το θέμα αυτό για τη χρηματοδότηση της υγείας. Φυσικά η προσέγγιση της ανακοίνωσής μας και των συμπερασμάτων του Συμβουλίου είναι κάπως ευρύτερες σε χαρακτήρα. Αυτό το οποίο θέλησαμε να κάνουμε εμείς στην Κομισιόν και νομίζω το ενστερνίστηκε και το Συμβούλιο είναι να θέσουμε τις δράσεις πολιτικής ανάπτυξης στο πλαίσιο μιας συνάφειας και συνοχής για εσωτερικά θέματα σημαντικά που, ενδιαφέρουν τις αναπτυσσόμενες χώρες, παραδείγματος χάρη το θέμα της μετανάστευσης με σαφή αποτελέσματα για την δύναμη εργασίας, τα ζητήματα επίσης εμπορίου, το θέμα της πρόσβασης στα φάρμακα, αλλά θέλουμε να εξασφαλίσουμε και την συνοχή με θέματα όπως είναι η επιστηστική ασφάλεια και το περιβάλλον. Ένα άλλο τομέα, ο οποίο ήταν ιδιαίτερα προεξάρχον σε αυτή την ανακοίνωση, ήταν το πώς η πολιτική ανάπτυξη μπορεί να συμβάλλει αποτελεσματικά σε μια οικουμενική κάλυψη στον υγειονομικό τομέα. Από την άποψη αυτή, δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην προσπάθεια να εξασφαλίσουμε και μεγαλύτερη ισοδικία στην κατανομή των βοηθειών μέσα στις διάφορες χώρες να έχουμε τη σωστή αρχιτεκτονική υγειονομική ε, περίθαλψη και να αντιμετωπίσουμε ιδίω τι ευάλωτε ομάδε του πληθυσμού, να ενισχύσουμε λοιπόν σε ασθενή κράτη στην υποσαχάρη Αφρική τα συστήματα υγειονομική περίθαλψη αλλά επίση και τα συστήματα σε άλλε χώρε του κόσμου. Πιστεύουμε ότι ο, ο κύριος τρόπος, ο καλύτερο τρόπο που μπορούμε να το κάνουμε είναι με την παροχή μεν βοήθειας η οποία είναι προβλέψιμη, σε οικονομικό επίπεδο αλλά και συγχρόνως με παράλληλες πολιτικές. Αυτό είναι κάτι το οποίο το είχε επισημάνει και το ελεγκτικό συνέδριο για την, στην έκθεσή του για την υγεία στην υποσαχάρια Αφρική. Μέσα σε αυτό το διάλογο βλέπουμε λοιπόν ότι μία από τις προτεραιότητες πρέπει να είναι η δίκαια χρηματοδότηση. Fair financing. Εργαζόμαστε πολύ για το θέμα αυτό από το 2009 μαζί με τους εμπλεκομένους ακαδημαϊκούς φορείς, ε, χώρες εταίρους και εδώ σίγουρα τίθεται ένα θέμα μεγάλης σημασίας. Η Κομισιόν <clears throat> δεν έχει μια συγκεκριμένη πολιτική γραμμή για την δίκαια χρηματοδότηση. Όπως ξέρετε, τα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν διαφορετικά συστήματα για την ε, χρηματοδότηση της υγειονομικής περίθαλψης. Θεωρούμε όμως ότι έχουμε κάποιες κοινέ αρχές για να μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε τη λειτουργία αυτών των συστημάτων που βασίζονται στην ποιότητα της ε, περίθαλψης, τον οικουμενικό της χαρακτήρα, την αλληλεγγύη και την εισοδική. Ένα από τα θέματα λοιπόν τα οποία πρέπει να κρατήσουμε στο μυαλό μας είναι το γεγονός ότι τα εθελοντικά συστήματα υγειονομικής ασφάλισης που αναφέρατε μπορεί να είναι πολύ ενδιαφέρουσες εμπειρίες σε πολλές χώρες, καλύπτουν ακόμα ένα πολύ μικρό ποσοστό των κατοίκων στην υποσαχάρια Αφρική το μισό περίπου της υγειονομικής περίθαλψης γίνεται από άμεσες πληρωμές των ασθενών προς τους ιατρούς και τα νοσοκομεία, κάτι το οποίο έχει πολλές φορές ένα πάρα πολύ σοβαρό αντίκτυπο στην, ε, στα νοικοκυριά, διότι είναι πάρα πολύ μεγάλες αυτές οι δαπάνες σε σχέση με τις οικονομικές δυνατότητες των νοικοκυριών και οδηγούν σε μεγαλύτερη ένδια. Λιγότερο από το 10% της ιδιωτικής δαπάνης για την υγεία περνάει μέσα από κοινά συστήματα όπως αυτά που αναφέρατε στις χώρες που παρακολουθήσαμε η κάλυψη της υγείας είναι αποσπασματική και εμβαλωματική και δεν φαίνεται να αυξάνεται ιδιαίτερα. Όπως είπατε και εσείς σωστά πρέπει να υπάρξει παράλληλα μια ενίσχυση των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης με εθνική αλλά και διεθνή υποστήριξη για χώρες οι οποίες έχουν μεγάλα προβλήματα στη χρηματοδότηση της δημόσιας υγείας. Εμείς προσβλέπουμε λοιπόν <clears throat> στην εξέταση της έκθεσης αυτής. Ελπίζουμε θα μπορέσουμε να συμμετάσχουμε και σε ανταλλαγή απόψεων σε μεταγενέστερες συνεδριάσεις και ελπίζουμε θα λάβει υπόψη την οικουμενική αυτή την παγκόσμια διάσταση υγείας. Πρέπει να υπάρχει οπωσδήποτε μια συνεκτική αντιμετώπιση με άλλες εσωτερικές πολιτικές και ένα άλλο σημείο όπου θεωρούμε ότι ίσως θα έπρεπε να το λάβει υπόψη στη συγγητρία είναι ότι αυτή τη στιγμή, όπως λέτε πολύ σωστά, υπάρχει μια πολλαπλότητα καθέτων πρωτοβουλειών, δηλαδή προγράμματα για ειδικέ ασθένειες. Έχουμε πάνω από 140 τέτοια προγράμματα και υπάρχει και κάποια σύγχυση σε εθνικό επίπεδο πολλές φορές σε σχέση με αυτές τις πρωτοβουλίες. Πολλές φορές οι κυβερνήσεις, οι υγειονομικοί φορείς και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δεν έχουν παίξει ένα πρωταρχικό ρόλο σε θέματα υγείας στην Ήπεθρο <clears throat> και πάρα πολλέ τέτοιε πρωτοβουλίε καλύπτονται από ιδιωτικού φορεί ή πολυμερει συμφωνίε. Λοιπόν, αυτέ είναι οι αρχικέ μα παρατηρήσει και προσβλέπουμε στη συνέχεια τη συζήτηση και στο να δούμε την ε, έγγραφη έκθεση της κυρία Ντεκέιζερ. Ευχαριστώ. Κυρία Ντεκέιζερ για τα συμπεράσματά της. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ τον κύριο Μίτσελ για τις αρχικές παρατηρήσεις του. Λυπάμαι που δεν έχει μεταφραστεί το κείμενο. Ευχαριστώ τον Σάλα και κυρίως αυτό που ανέφερε για την ε, περιφερειακή διάσταση. Θα το δω αυτό και θα την ε, εντάξει αυτή την ιδέα στο κείμενό μου, στην έκθεσή μου. Είναι μια διάσταση η οποία όντως πολύ σωστή σε σχέση με τους στόχους της εκθέσεως. Ευχαριστώ και την Επιτροπή για όλες τα σχόλια. Φυσικά έλαβα υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, τις συστάσεις του Ελεκτικού Συνεδρίου εννοείται. Ευχαριστώ για όλα θα δούμε πώς μπορώ όλα αυτά να τα διαρθρώσω, να τα ενσωματώσω. Αλλά να απλώς να πω ότι μια έκθεση πρωτοβουλίας δεν έχει σαν στόχο να επαναλάβει όλα αυτά τα συμπεράσματα τα οποία έχουν επιτευχθεί. Ε, έτσι δεν δημιουργείται θέμενη αξία. Ε, ο στόχος είναι φυσικά στα σωστά πλαίσια να θίξει κάποια σημεία, τα σημεία τα οποία εγώ θεωρώ ότι πρέπει να υπογραμμίσουμε. Εννοείται, ε, ε η ιδέα δεν είναι να ξανασυντάξουμε, να κάνουμε μια προσαρμογή κειμένων που ήδη υπάρχουν. Με αυτές τις λίγες παρατηρήσεις θα φύγω εγώ τώρα και Επίσης υπάρχει και ένα σημείο το οποίο έχει να κάνει με το ταξίδι που κάναμε στη Γάζα, ένα από εκείνο ταξίδι και στην Παλαιστίνη, στο Ισραήλ. Δυστυχώς δεν θα μπορώ να είμαι παρούσα όταν θα δείτε αυτό το κείμενο. Ε, θα μας λείψετε λέει η πρόεδρος. Περνάμε στο σημείο 8. Παρακολούθηση της δημοσιονομικής στήριξη στις ανεπτυσσόμενε χώρε. Όπως ήδη ξέρετε, η Επιτροπή Ανάπτυξης ζήτησε μια μελέτη για εντοπίσει κανείς ε, το βαθμό αποτελεσματικότητας του κοινοβουλευτικού ε, όσον αφορά το, τους προπολογισμούς στις ε, χώρες εταίρους. Επίσης, έχει γίνει αναλύσεις και βλέπει κανείς πώς ε, για την Πουρκίνα Φάσο Γκάνα τη Δημοκρατική Δρομοκρατία να δει ε, κατά επιθυμία του ελεκτικού συνεδρίου να δει κανείς πώς ακριβώς ε, έχουν τα πράγματα. Θα δώσω τώρα το λόγο της συγκυρία Σβέα Κοχ, εκπρόσωπος του Ινστιτούτου Σίτβιτ, να μας ενημερώσει. 20 λεπτά θα έχει στη διάθεσή της. Um, Ευχαριστώ. Καλό απόγευμα. Νομίζω ότι πρέπει να δούμε τέσσερα ερευνητικά ερωτήματα τα οποία έχουν διατυπωθεί και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Καταρχήν ο ρόλο των κοινοβουλίων και αποτελεσματικότητα στην παρακολούθηση τη υποστήριξη του προπολογισμού. Δεύτερον, ο ρόλο και η αποτελεσματικότητα των ελεκτικών φορέων σε ό,τι αφορά την παρακολούθηση τη βοήθεια προ τον προπολογισμό. Τρίτον, το βαθμό κατά τον οποίο οι αποφάσει των χορηγών για τον προπολογισμό υπόκεινται στην εξέταση των εθνικών μηχανισμών ελέγχου. Και τέταρτον, το, η έκταση και αποτελεσματικότητα των εξαρτήσεων και των συμπληρωματικών μέτρων για να βελτιωθούν οι εθνικοί μηχανισμοί ελέγχου. Τα στοιχεία μας τα έχουμε συλλέξει από συνεντεύξεις σε τρεις χώρες, Γκάνα, Μπουρκίνα Φάσο και Δομινικανική Δημοκρατία. Παρά το γεγονό ότι φαίνεται ότι είναι καλή η απόδοση στι περιπτώσει αυτέ, υπάρχουν σημαντικέ ελλείψει στου εθνικού ελεγκτικού μηχανισμού. Και η πολιτική κατάσταση, οι μηχανισμοί ελέγχου διαφέρουν τα μάλα. Οι χώρε αυτέ αποτελούν μια καλή βάση σύγκριση περιπτώσεων όπου η υποστήριξη αποτελεί ένα μεγάλο μέρο του εθνικού προπολογισμού, Παραδείγματο χάρη στην Μπουρκίνα Φάσο, στην Γκάνα είναι 30% και η αντίθετη περίπτωση είναι ενό ασήμαντου υπο, ποσοστού υποστήριξης 4% στη Δομινικανική Δημοκρατία. Για τα κοινοβούλια. Η υποστήριξη του προπολογισμού συγχαίρεται πλήρω με, τον εθνικό κοινο, με εθνικό προπολογισμό, θα πρέπει να υπάρξει μια αξιολόγηση στα πλαίσια του σύνολου προπολογισμού και δεν παραμένει μονάχα στα επίπεδα τη υπόσταση. Βλέπουμε όλο τον προπολογισμό λοιπόν και το συνολικό ρόλο των κοινοβουλίων εξάντε εξ Οι πελέτες δείχνουν ότι ο συνολικό ρόλο των κοινοβουλίων σε όλε τι αυτέ τι χώρε είναι ασθενή λόγω του γεγονότο, ότι υπάρχουν πολλέ μορφέ περιορισμών σε θεσμικό και διοικητικό επίπεδο και είναι πολύ λίγε οι ενδείξει ότι έχει βελτιωθεί η λειτουργία του λόγω τη υποστήριξης των προπολογισμών. Έχουμε δύο θετικά παραδείγματα, καταρχήν στην περίπτωση τη Γκάνα στο επίπεδο ex post υπήρξε μια μεγαλύτερη οκίτητα σε ό,τι αφορά τον δημόσιο έλεγχο και την ε, εξέταση από δημόσιες ε, ε, επιτροπές με δημόσιες ακροάσεις επίσης υπήρξε σημαντική βελτίωση και επίσης τη δομινικανική δημοκρατία σε ό,τι αφορά την αποτελεσματικότητα έχουν τώρα νέους φορείς που δίνουν την δυνατότητα στο κοινοβούλιο τους να αντιμετωπίσει τον προϋπολογισμό εγκαίρως και να έχει ένα καλύτερο πλαίσιο. Είδαμε επίσης ότι τα κοινοβούλια δεν ενσωματώνονται πλήρως στη διαδικασία υποστήριξη του προϋπολογισμού. Παραδείγματο χάρη με ετήσιες ε, εξετάσεις ή με δυνατότητα διαλόγου. Στον Μπουρκίνα Φάσου ζητήθηκε κάτι τέτοιο να γίνει, αλλά υπήρξε μια αντίρρηση από ορισμένους χορηγούς. Στις ε, ανταλλαγές απόψεων με την Κομισιόν μάθαμε ότι οι κοινοβουλευτικοί στον Μπουρκίνα Φάσο προσεκλήθησαν ως παρατηρητές να συμμετάσχουν στο διάλογο πολιτικής αλλά όλοι οι κοινοβουλευτικοί που είδαμε δεν ξέραν όλοι ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Αυτό δείχνει ότι η ροή πληροφοριών είναι ανεπαρκής. Γι' αυτό στην Κάνα παραδείγματος χάρη και στη Δομινικανική Δημοκρατία είδαμε πάρα πολλοί κοινοβουλευτικοί να μην ξέρουν τίποτα ότι υπάρχει υποστήριξη του προπολογισμού. Στην Πουρκίνα Φάσο οι κοινοβουλευτικοί πρέπει να εγκρίνουν όλες τις συμφωνίες για δάνεια, αλλά δεν έχουν πλήρη πληροφόρηση. Συνολικά λοιπόν η βοήθεια στον προϋπολογισμό είναι σημαντική για να υπάρξει καλύτερη μορφή ελέγχου των μορφών βοήθειας από τα κοινοβούλια, αλλά αυτό δεν ενισχύει το ρόλο των κοινοβουλίων εάν δεν υπάρχει μια εναρμονισμένη δράση των ε, χορηγών που να περιλαμβάνει και τα κοινοβούλια. Σε ό,τι αφορά τα ανώτατα ελεκτικά όργανα, είδαμε ότι μετά από την εισαγωγή της υποστήριξης στο προπολογισμό, οι θεσμοί και, στους και στις τρεις χώρες ενισχύθηκαν. Στη Δομινικανική Δημοκρατία έχει αυξηθεί σημαντικά η ανεξαρτησία του ελεκτικού συνεδρίου και είναι το κοινοβούλιο που διορίζει τα μέλη του ελεκτικού συνεδρίου, ενώ προηγουμένως ήταν ο πρόεδρος της χώρας. Επίσης και στην Μπουρκίνα Φάσο και στην Γκάνα έχει βελτιωθεί η κατάσταση. Στην Γκάνα η έκθεση για το 2008 ήταν η πρώτη φορά που υπευλήθη στο Κοινοβούλιο μέσα στο, στην ε, προβλεπόμενη προθεσμία 6 μηνών ενώ μέχρι το 2007 συζητούσαν εκθέσει τρία χρόνια πίσω. Η κύρια πρόκληση είναι να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα του ελεκτικού χαρακτήρα των θεσμών αυτών. Όπως είδαμε σε ό,τι αφορά το Κοινοβούλιο, επίσης και οι ανώτατοι ελεκτικοί φορείς δεν ενσωματώνονται πλήρως στη διαδικασία υποστήριξη του προϋπολογισμού. Στις ε, περιπτώσεις που είδαμε δεν έχουν πραγματικά πολλά στοιχεία για τις ε, ροές βοήθειας, Πραγματικά χάρη στη Δομινικανική Δημοκρατία. Είδαμε ότι δεν χρησιμοποιεί το πλήρως το έγγραφο που παρουσίαζε τι χρηματικέ ροές και είναι πολύ άσχημα πληροφορημένη σε σχέση με την υποστήριξη προς τον προπολογισμό. Σε σχέση με το δεύτερο στόχο της δήλωσης του Παρισίου, είδαμε ότι υπάρχει καλύτερη λειτουργία των εθνικών συστημάτων ελέγχου και μείωση των παράλληλων μηχανισμών. Αυτό όμω έχει να κάνει και με την ικανότητα των εθνικών μηχανισμών ε, ελέγχου αυτό γίνεται παραδείγματος χάρη σε χώρε όπω η Γκάνα, αλλά όχι στη Δομινικανική Δημοκρατία. Για τους εσωτερικούς φορείς φαίνεται ότι δεν υποστηρίζονται τόσο πολύ από τους χορηγούς όσο τα ανώτατα ελεκτικά εδρήματα θεωρούνται γενικά ότι είναι πολύ κοντά στο κράτος και αυτό δεν τους δίνει δυνατότητα να δράσουν ως ανεξάρτητοι μηχανισμοί ελέγχου. Κοιτάξαμε επίση του εμπλεκόμενου από την κοινωνία των πολιτών, ιδίω σε χώρε όπου είναι ασθενεί η διαχείριση των δημοσίων οικονομικών έχουν να παίξουν ένα σημαντικό συμπληρωματικό ρόλο. Είδαμε σε όλε αυτέ τις χώρε ότι τα μέσα ενημέρωση και μη κυβερνητικοί οργανισμοί ενισχύουν ιδιαίτερα την έλεγχο του προπολογισμού και δημιουργούν ένα κλίμα όπου οι φορεί εφαρμογή του προπολογισμού είναι πιο υπόλογοι. Η βελτίωση των εθνικών μηχανισμών ελέγχου και η ανάπτυξη ενός συστήματος λογοδοσίας σε εθνικό επίπεδο βασίζονται και στην ενισχύση της λειτουργίας και της συμμετοχής του Κοινοβουλίου, όπως φάνηκε αυτό στην περίπτωση της Γκάνας. Υπάρχει λοιπόν και μεγαλύτερη επίγνωση για τα θέματα αυτά από την πλευρά των πολιτών. Πρέπει να ενισχύσουμε λοιπόν αυτή την συνέργεια που μπορεί να υπάρχει. Για το τρίτο ερώτημα για την αξιολόγηση από την πλευρά των χορηγών των εθνικών μηχανισμών ελέγχου το, η αξιολόγηση PIFA, κανείς δεν ξέρει εδώ πέρα μάλλον τι είναι η PIFA, η PIFA έχει αναπτυχθεί από τους δωρητές για να υπάρχει ένα κοινό πλαίσιο δημοσιονομικής διαχείρισης και υπήρξε και μία αξιολόγηση και στις τρεις χώρες που ανέφερα. Το γεγονός ότι τα κοινοβούλια και οι ελεκτικοί φορείς δεν πέτυχαν υψηλή βαθμολογία, αυτό δεν είχε κανένα αποτέλεσμα. Στην περίπτωση της Δομινικανικής Δημοκρατίας πήραν όλοι οι φορείς στο χαμηλότερο δυνατό βαθμό. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χρησιμοποιεί μια δυναμική ερμηνεία επιλεξιμότητος. Θεωρεί ότι ακόμα και χώρες όπου η δημόσια διαχείριση των οικονομικών είναι ασθενής, αυτό δεν τις αποκλεί από την παροχή υποστήριξης για τον προϋπολογισμό, γιατί ο στόχος είναι να υπάρξει μια καλύτερη μεταρρύθμιση και εφαρμογή δεν υπάρχει και καμία άμεση σχέση μεταξύ των αποτελεσμάτων αυτής της αξιολόγησης και της επιλεξιμότητας για υποστήριξη στον προϋπολογισμό. Ο στόχος είναι περισσότερο να προωθηθεί η μεταρρύθμιση και όχι να βελτιωθεί η πραγματική κατάσταση. Γενικά λοιπόν οι κατευθυντήριες γραμμές δεν οδηγούν σε μια υποχρεωτική εξέταση των εθνικών μηχανισμών. Και ο ορισμός του τι είναι εθνικός μηχανισμός είναι κάπως ανεπαρκής γιατί δεν περιλαμβάνει πάντα τους εμπλεκόμενους στην κοινωνία των πολιτών, το κοινοβούλιο και τα ανώτατα ελεκτικά ιδρύματα. Αν δούμε λοιπόν τον κύκλο λογοδοσίας, αν δούμε την ε, ε, διαδικασία, οι χορηγοί εστιάζουν περισσότερο στην εσωτερική, στον εσωτερικό κύκλο, την ε, αν θέλετε, κεντρική διαδικασία, ενώ οι εμπλεκόμενοι στην κοινωνία των πολιτών που βρίσκονται στον εξωτερικό ομόκυδο κύκλο δεν λαμβάνονται τόσο υπόψη. Για το τέταρτο ερευνητικό ερώτημα, την εξαρτησιμότητα και τους μηχανισμούς ελέγχου, η διαδικασία διαχείρισης με στο πλαίσιο που ανέφερα είναι κάτι πολύ σημαντικό για τους χορηγούς σε όλες τις χώρες αυτές και οι εξαρτήσεις καθώς και τα συνοδευτικά μέτρα είχαν θετικά αποτελέσματα στην διαχείριση των ε, οικονομικών. Οι χορηγοί σε κάποιο βαθμό έχουν προσπαθήσει να βελτιώσουν τη δημιουργία ικανότητα στα κοινοβούλια αλλά επίσης και στους ανώτατους του ΣΥΠΑ, τους ελεκτικούς φορείς, κάτι το οποίο βοήθησε σε μια καλύτερη λειτουργία των θεσμών αυτών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι στιγμή δεν έχει πετύχει πολλά σε επίπεδο ενίσχυσης των κοινοβουλίων. Είναι περισσότερο σημαντικό οργανισμό τη Παγκόσμια Τράπεζα του Καναδικού Κέντρου για την Ενίσχυση των Κοινοβουλίων, αλλά όχι τη Κομισιόν. Είδαμε ότι η χρηματοδότηση του προπολογισμού και τα μέτρα που τα συνοδεύουν δεν είναι απόλυτα ισορροπημένα. Στην περίπτωση της Δομικανικής Δημοκρατίας και της Πουρκίνο Φάσο δεν υπήρξε χρηματοδότηση για την χρηματοδότηση μηχανισμών έλεγχου. Ενώ για το έγγραφο στρατηγικής της Κάνα 2% του προγράμματος είχε σαν στόχο να υποστηρίξει τους φορεί της κοινωνίας των πολιτών που μπορούν να είναι οι ελεγκτές και οι παρατηρητές αυτών των θεμάτων. Αυτό δεν γίνεται όμως με συστηματικό τρόπο ακόμα. Και στην περίπτωση ακόμα της Γκάνα, ακόμα και αν αυτό είναι κάτι το οποίο είναι θετικό, χρειάζεται και εκεί μια βελτίωση της χρηματοδότησης. Εν γέννη, καταλήξαμε στο ότι είναι μικρή η υποστήριξη που δίνεται από τα μέτρα αυτά για ενίσχυση του προϋπολογισμού στο σύστημα εσωτερικής ε, λογοδοσίας. Βασικά, η λογοδοσία αυτή εστιάζεται σε τεχνικές και διοικητικές πτυχές, ενώ η ενίσχυση του Κοινοβουλίου των Ανεξαρτήτων Μέσων Ενημέρωσης και της κοινωνίας των πολιτών πρέπει να παίξει ένα σημαντικό ρόλο. Πρέπει να ενισχύσουμε λοιπόν την εσωτερική λογοδοσία και πρέπει να τονίσουμε ότι με την ενίσχυση του προπολογισμού αυτό δεν επιτυγχάνεται ε, αυτόνομα χωρίς να υπάρξει μια πραγματική αλλαγή μέσα στον εσωτερικό πολιτικό ιστό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό σε χώρες όπως η Μπουρκίνα Φάσο. Πρέπει να υπάρχει όμως και μια δέσμευση των χορηγών για να ενισχυθούν αυτοί οι μηχανισμοί ελέγχου για να μπορέσουμε να ενισχύσουμε την υποστήριξη των μηχανισμών αυτών σε μακροπρόθεσμο επίπεδο. πέντε κύριες συστάσεις από τη δική μας πλευρά. Καταρχήν, στον προγραμματισμό, το σχεδιασμό και την εφαρμογή της υποστήριξης του προπολογισμού θα πρέπει να υπάρχει μια σαφής και ολιστική αντιμετώπιση των μηχανισμών ελέγχου. Θα πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον δύο μορφή λογοδοσία και οριζόντια και διασταυρούμενη έλεγχη μέσα στη χώρα αυτή και η ικανότητα των κρατικών φορέων να εγκαλούν την κυβέρνηση και να την ελέγχουν, αλλά υπάρχει και μια άλλη μορφή λογοδοσίας, η κάθετη λογοδοσία που είναι οι μηχανισμοί των φορέων της κοινωνίας των πολιτών για να ελέγξουν την κυβέρνηση. Είναι απαραίτητο να δούμε ότι το Κοινοβούλιο παίζει σημαντικό ρόλο και στις δύο μορφές λογοδοσίας, στη μία πλευρά την κάθετη είναι και οι εκπρόσωποι των πολιτών. Δεύτερη σύσταση, οι εμπλεκόμενοι για τους, οι εμπλεκόμενοι στον Εθνικό Μηχανισμό Ελέγχου, όπως τα κοινοβούλια, θα πρέπει να τύχουν καλύτερες αξιολόγησεις πριν από την παροχή άμεσης υποστήριξης και ζητούμε να υπάρξει μια καλύτερη παρακολούθηση και έλεγχος των κοινοβουλίων, να δούμε και ποια είναι η απόδοση και η λειτουργία των κοινοβουλίων, για να δούμε αν είναι σε θέση να μπορέσουν να παίξουν αυτό το ρόλο και να δούμε ποιε είναι και οι εξωτερικές αδυναμίες για το θέμα αυτό. Χρειάζεται λοιπόν μια πλήρης αξιολόγηση τη ικανότητα των κοινοβουλίων κατά περίπτωση. Αν δείτε πού είναι τα ισχυρά και τα ασθενή σημεία, μπορεί κανεί να έχει μια εναρμονισμένη προσέγγιση για να δούμε πώ ο κάθε χορηγό μπορεί να αντιμετωπίσει τα προβλήματα αυτά. Και σα λέω ότι αυτό θα πρέπει να γίνεται με την ε, πρωτοβουλία των ίδιων χωρών. Είναι σημαντικό επίση να παρακολουθούμε την ε, λειτουργία των κοινοβουλευτικών φορέων για να δούμε ποιοι είναι οι κίνδυνοι και η αποτελεσματικότητα των ελέγχων και επίση να παρακολουθήσουμε και τα αποτελέσματα τη ανάπτυξη ικανότητα. Επίση, η Κομισιόν θα πρέπει να εξασφαλίσει καλύτερη υποστήριξη της ε, υποστήριξης του προπολογισμού και τη ανάπτυξη κερίων θεσμών που μπορούν να είναι οι εθνικοί φορεί ελέγχου. Επειδή αυτοί οι φορεί μπορεί να είναι μη αποτελεσματικοί σε ορισμένε χώρε, ένα ποσοστό της ε, υποστήριξη του προπολογισμού θα πρέπει να προσδιορίζεται αποκλειστικά για την, για την ενίσχυση της <clears throat> λογοδοσίας και της λειτουργίας αυτών των φορέων με τη συμμετοχή των κοινοβουλίων στο πλαίσιο αυτό θα μπορούσε να προκύψει μια βελτίωση. Αλλά θα πρέπει να ξέρουμε ότι θα πρέπει να υπάρχει και έλεγχος από τις εκτελεστικές αρχές σε σχέση με τους ε, ενδείκτες για την επίτευξη των στόχων. Αυτό είναι πολύ σημαντικό λοιπόν σε ό,τι αφορά την έγκαιρη υποβολή του προπολογισμού στο Κοινοβούλιο, αλλά αυτό πρέπει να το εξετάσουμε αναχώρα. Πιστεύω ότι το πιο εφικτό είναι αυτή τη στιγμή να ενσωματωθούν και τα κοινοβούλια και η φόρηση, η ανώτατη ελεκτική φόρεις στη διαδικασία ελέγχου των ροών προς τον προπολογισμό, αλλά πρέπει να γίνει αυτό όχι με επιλογή τυχαίων κοινοβουλευτικών, αλλά με κοινοβουλευτικού οι οποίοι εμπλέκονται στην Επιτροπή Οικονομικών και Δημοσίων Οικονομικών των χωρών αυτών για να μπορούν αυτοί να παρακολουθούν τα τεκτενόμενα και να κάνουν μια έκθεση στο Κοινοβούλιο. Εάν δεν υπάρχει θέληση της κυβέρνησης θα μπορούσαν να υπάρχουν αιτήσει ή ανά δύο έτη εκθέσεις προς το Κοινοβούλιο που να καλύπτουν όλα τα στοιχεία τα οποία έχουν τύχει συμφωνία στον πολιτικό διάλογο ώστε το Κοινοβούλιο της κάθε χώρας να ξέρει τι ακριβώ έχει αποφασιστεί. Μια πρόσφατη εξέλιξη στην Κάνα είναι ότι έχουν ξεκινήσει μια κοινοβουλευτική πλατφόρμα για την πολυμερή, πολυμερή υποστήριξη προς το υπολογισμό για να έρθουν οι κοινοβουλευτικοί και οι χορηγοί καλύτερα μεταξύ τους να συζητούν για τα θέματα του, των στόχων της χιλιετίας και να έχουν μια ευρύτερη βάση υποστήριξη. Αυτό είναι ένα πολύ θετικό βήμα, αλλά είναι πολύ νωρί να πει κανείς αν αυτό το μέτρο θα είναι θετικό ή όχι. Η συστάση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να περιλάβει το θέμα της υποστήριξης του προπολογισμού και της παρακολούθησης του κοινοβουλευτικού προπολογισμού στο διάλογο με χώρες Ακέ στα πλαίσια της ε, ε, Μικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ευρωπαϊκή Ένωση και, και μέσα στην βοήθεια του Γραφείου για την προώθηση της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Επίσης βλέπουμε ότι η Κομισιόν αναθεωρεί τις καταθυντήρες γραμμές της και η πράσινη βίβλος για την υποστήριξη του προπολογισμού θα διατυπωθεί αυτό το φθινόπωρο. Επομένως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι όλες αυτές οι συστάσεις περιλαμβάνονται στην πράσινη αυτή βίβλο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Γκέρεν, ζητήσατε το λόγο. θεωρώ πολύ χρήσιμη αυτήν την προσέγγιση. Θα ήθελα όμως να ξέρω ποια θα είναι η συνέχεια. Αν ήσασταν στη θέση της Επιτροπής που θα διαπραγματευτεί αυτές τις ε, συμφωνίες για υποστήριξη όσον αφορά το υπερπολογισμό. Θα είχατε μια προσέγγιση αυστηρή. Αυτό σαν μια ερώτηση. Το δεύτερο έχει να κάνει με τη διαφθορά. Ξέρετε ένα έστω παράδειγμα όπου έχετε, έχετε ικανοποιητική κατάσταση εκτέλεση όσον αφορά ε, την εκτέλεση του προπολογισμού και όπου είναι κακοπληρωμένοι οι, οι υπάλληλοι, οι δημόσιοι υπάλληλοι. Θα μπορούσατε να μας πείτε αν μπορεί κανείς να πετύχει όντως μια σωστή, σωστή χρηστή, χρηστή διαχείριση του προπαλογισμού. Ε, συχνά, ε, συχνά δέχεται κανείς ε, ανόητες ίσως ε, θα λέγαμε ερωτήσεις και εγώ να το κάνω και εγώ με το δικό μου τρόπο. Ευχαριστώ. Κρίμα που δεν ήμουν παρούσα. Ζητώ συγγνώμη για το πρώτο τμήμα τη παρουσίασή σα. Ήμουν σε μια άλλη συνεδρία. Βλέπουν την έκθεσή σα ή το σχέδιό σα τη έκθεση υπάρχουν δύο στοιχεία τα οποία δεν είναι πολύ σαφή για μένα. Καταρχήν, ποιο είναι το ποσοστό που υποστήριξη του προπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, <clears throat> του προπολογισμού των χωρών στι οποίες κάνατε την έρευνά σα, και αναρωτιέμαι αν υπάρχουν στατιστικέ που δείχνουν αύξηση ή μείωση της υποστήριξης του προπολογισμού στις χώρες που μελετήσατε. Και αυτό θα είναι ενδιαφέρον να το παρακολουθήσει Κανεί. Και έχουν χάσει το πρώτο τμήμα της παρουσίασή σα, Ίσως θα θέσω ένα ηλίθιο ερώτημα, αλλά ίσως είναι ενδιαφέρον παρόλα αυτά. Τι θα λέγατε από την εμπειρία σας στις χώρες αυτές τις οποίες κοιτάξατε, τι είναι αυτό που κάνει τα κοινοβούλια καλύτερα ικανά να ελέγξουν τα οικονομικά. Γιατί τα κοινοβούλια σε καλύτερη θέση να προχωρήσουν σε αυτό τον έλεγχο. Έχετε κάνει ορισμένε συστάσει, αλλά τι είναι αυτά τα οποία έχουν λειτουργήσει καλά στο παρελθόν και τι είναι αυτά τα οποία δεν λειτουργήσαν καλά στο παρελθόν. Ευχαριστώ. Κύριο äh, um- Ευχαριστώ για αυτή την πλήρη έκθεσή σας. Νομίζω ότι αυτή η έκθεση είναι απόλυτα σημαντική και χρήσιμη, <clears throat> γιατί εμείς συζητούμε για την αναπτυξιακή βοήθεια και με τους πολίτες μας πάντα θέλουμε να ανταποκριθούμε στο αίτημα των πολιτών μας για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Και η έκθεση έχει αυτή πάρα πολλά σημεία, τα οποία θέτουν τον δάκτυλο επί τον τύπο των ύλων της αποτελεσματικότητας αυτής της υποστήριξης προς τον προϋπολογισμό. Σίγουρα η υποστήριξη προς τον προπολογισμό είναι πάρα πολύ σημαντική για να μπορέσει να ενισχύσει και να εξελίξει περαιτέρω τις κοινοβουλευτικές δομές στις χώρες αυτές. Αλλά επειδή έχετε απλώς αυτήν την προσωρινότητα στην έκθεσή σας, νομίζω ότι εμείς θα πρέπει να έχουμε και σαφέστερες ενδείξεις για το πώς γίνεται ο έλεγχος από την πλευρά της και επίσης πώ μπορούμε εμεί ω κοινοβουλευτικοί να ελέγξουμε την Κομισιόν σε ό,τι αφορά τον έλεγχο αυτό. Νομίζω ότι αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά στοιχεία τη κοινή μα εργασία. Η Κομισιόν, δεν ξέρω ποιο έχει το λόγο από την πλευρά τη Κομισιόν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ονομάζομαι Ζωζέ Κοριαλούνες, είμαι τμηματάρχη της γενική διεύθυνση που ασχολείται με την οικονομική στήριξη και την οικονομική διακυβέρνηση ε, μαζί με τον συνάδελφο Μάικ Φορμαντίνη βρίσκομαι εδώ από την ΕΚΟ που είναι εδώ και θα έχει την ευκαιρία και εκείνος να μιλήσει. Καταρχήν ευχαριστώ τους συντάκτες της μελέτης. Ε, είναι μια μελέτη πολύ καλή, πολύ ποιοτική. Το περιεχόμενο και τα στοιχεία είναι σωστά. είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε με τους συντάκτες της μελέτης και να ανταλλάξουμε ιδέες και πιστεύω πως είμαστε στη καλή πορεία. Όπως είπε και όλας η κυρία που έκανε την εισήγηση, η Κομισιόν αυτή τη στιγμή σκέφτεται το θέμα της οικονομικής στήριξης όχι μόνο μέσα στο πλαίσιο της βελτίωσης ε, του ίδιου του μέσου, αλλά και με βάση τους διάφορους ε, φορείς που συμμετέχουν όπως το Κοινοβούλιο, τα όργανα ελέγχου και η κοινωνία των πολιτών. Και οι δράσει μας περιλαμβάνουν διάφορους ε, πυλώνε. Καταρχήν, και αυτό αναφέρθηκε, υπάρχουν εργασίε για τη βελτίωση του οδηγού για την δημοσιονομική στήριξη. Είναι αλήθεια και αυτό το διαπιστώνουμε ότι αν και αναφέρεται το Κοινοβούλιο, το χώρος που υπάρχει αυτό δεν είναι αρκετά μεγάλος, άρα τα θεσμικά όργανα που είναι υπεύθυνα για την παρακολούθηση και την έλεγχο. Δεν αναφέρονται παρκώ σε αυτό. Ε, προσπαθούμε να το διορθώσουμε ώστε να καταλάβουμε τις διάφορες πτυχές νομιμότητας όσον αφορά την δημοσιονομική στήριξη συμπεριλαμβανομένες δημόσια οικονομία, αλλά και όλων των φορέων που εμπλέκονται όχι μόνο της κυβέρνησης αλλά και των υπολείπων στο πλαίσιο του διαλόγου που έχουμε με τις ε, χώρες δικαιούχους. Ένα άλλο άξονα είναι φυσικά ο προβληματισμός γύρω από ένα πράσινο βιβλίο και εκεί πιστεύω πως είναι η θα είναι η ευκαιρία για να συζητήσουμε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να λάβουμε υπόψη τις ε, συστάσεις ε, της έκθεσης και για να ενσωματωθούν όλα αυτά στην δημόσια συζήτηση που θα γίνει πιστεύουμε στα μέσα του έτους, δηλαδή από τη στιγμή που θα έχει ε, ξεκινήσει το πράσινο βιβλίο. Δηλαδή, πράσινο βιβλίο σημαίνει εντοπισμό των θεμάτων που θα πρέπει να εξεταστούν. Και σας διαβεβαιώ πως ε, ε, όλα αυτά θα συμπεριλαμβάνονται στο πράσινο βιβλίο και η συζήτηση θα ξεκινήσει Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Ελπίζω. Για την ίδια την έκθεση, όπως σας είπα, είναι πολύ καλή, τα στοιχεία είναι σωστά, αλλά Είμαστε ανοιχτοί να συνεχίσουμε τη συζήτηση με του συντάκτε, γιατί κρίνουμε πω υπάρχουν ορισμένε πτυχέ που θα πρέπει να ε, τι ξαναδούμε, επί τη βάση δηλαδή των στοιχείων που μπορούμε να δώσουμε στου συντάκτε. Για παράδειγμα, όταν μιλάμε για την στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς ε, του ελεγκτικού οργανισμού, Οι συνάδελφοι τη ΕΚΟ μπορούν να δώσουν στοιχεία να δώσουν άλλο ένα πράγμα είναι τα ποσά και ένα άλλο πράγμα είναι η ορατότητα αυτών των κονδυλίων που δεν συμβαδίζουν πάντοτε. Και το σημαντικότερο θέμα που θέλω εγώ να θίξω εδώ είναι το θέμα της οικονομικής διακυβέρνησης και της πολιτικής διακυβέρνησης. Η έκθεση θίγει τις πτυχές της οικονομικής διακυβέρνησης, το ρόλο δηλαδή των κοινοβουλίων σε αυτή τη διακυβέρνηση που είναι πολύ σημαντικός. Αλλά χωρί σωστή διακυβέρνηση πολιτική, χωρί θεσμού που να λειτουργούν σε ένα δημοκρατικό πλαίσιο, αυτή η οικονομική διακυβέρνηση δεν πρόκειται να συμβεί. Άρα είναι αλήθεια ότι χρειάζεται να στηριχθούν τα κοινοβούλια στον ρόλο τους ε, ώστε να, κάνουν, ε, να παρακολουθούν και να ελέγχουν τον την εκτέλεση του προπολογισμού, αλλά τα κοινοβούλια αυτά θα πρέπει να αναγνωρίζονται από τους άλλους κρατικούς θεσμούς. Αυτό είναι πολύ σημαντική πτυχή της συζήτησης που κάνουμε με τους εταίρους αλλά και με τα κράτη-μέλη. Δηλαδή, το θέμα της οικονομικής στήριξης που εμείς εστιάζουμε στην οικονομική διακυβέρνηση και από την άλλη πλευρά τα ζητήματα που προκύπτουν τώρα από τη συζήτηση και αφορούν το πολιτικό, την πολιτική πτυχή και κυρίως τις βασικές αρχές που εντάσσονται στο πλαίσιο της εταιρική μας σχέση, είτε είναι η είτε είναι άλλες εταιρικέ σχέσεις. Είναι βασικές αξίες δηλαδή, κράτος δικαίου, δημοκρατία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το ένα μπορεί να ενισχύσει το άλλο, αλλά εργαζόμαστε σε ένα πλαίσιο και για ορισμένε χώρε που δεν θέλω τώρα να αναφέρω, όπου ανέλησαν οι συντάκτες, υπάρχουν προβλήματα σημαντικά όσον αφορά την πολιτική διακυβέρνηση. Αυτή είναι μια πτυχή που θα πρέπει να τη συζητήσουμε στο πλαίσιο της δημοσιονομικής στήριξης, γνωρίζοντα ότι η, οικονομική, η πολιτική διακυβέρνηση δεν θα γίνει ξαφνικά αλλά περισσότερο μέσα στο πλαίσιο πολιτικής, πολιτικού διολαού, μέσα στο πλαίσιο της Συμφωνίας Κοτονού, ας πούμε, στο, από το άρθρο 8, όπου πρέπει να ενισχυθεί ο πολιτικός διάλογος και στο πλαίσιο των υπολείπων εταιρικών ε, σχέσεων. Άλλη σημαντική πτυχή που ίσως θα μπορέσουμε αργότερα να συζητήσουμε τις τεχνικές της πτυχές είναι, το επίπεδο, είναι στο επίπεδο των συστάσεων. Είναι αλήθεια ότι η προσέγγιση μας είναι ότι θα πρέπει να κάνουμε έναν διάλογο που θα καλύπτει θα περιλαμβάνει τα Εθνικά Κοινοβούλια, την κοινωνία των πολιτών και το ελεγκτικά, τους ελεγκτικούς αλλά θα πρέπει πάντα να προσέχουμε ώστε τα Εθνικά Κοινοβούλια να μην πάρουν τη θέση ενός παρατηρητή σε μια, έναν διάλογο με την κυβέρνηση, όπου έχουν περισσότερο παθητικό ρόλο. Το παράδειγμα της Γκάνα δεν το γνωρίζω γιατί είναι καινούριο, αλλά θα έπρεπε να συμβαίνει το αντίθετο. Το Εθνικό Κοινοβούλιο να μπορεί να καλέσει τους δωρητές ώστε να συζητήσει μαζί τους και να έχει την αρχηγική θέση, την πρωτοπόρα θέση και μέσα σε αυτό το πλαίσιο να μπορέσουμε να εργαστούμε γιατί διαφορετικά βεβαίως στο πλαίσιο του διαλόγου με το εκτελεστικό σώμα αυτό καθοδηγεί την συζήτηση και το διάλογο, δηλαδή η κυβέρνηση. Πρέπει να λάβουμε υπόψη λοιπόν τις εξουσίες των μεν και των δε. Άλλη πτυχή είναι αυτή το επίδομα 3 με 5%. Από την εμπειρία μας βλέπουμε ότι αν δώσουμε συγκεκριμένα κονδύλια σε, κάποιο μόνο συγκεκριμένο τομέα, αυτό μπορεί να έχει αντίστροφα αποτελέσματα. Στη συζήτηση, γιατί γνωρίζουμε ότι οι προπολογισμοί είναι διαιτησίες. Διαιτησίες ανάμεσα στους υπουργούς, ανάμεσα στα υπουργεία, πολιτικές ε, ε, ρυθμίσεις και συχνά ε, συμβαίνει ο δωρητής να προσπαθεί να εξασφαλίσει ένα Υπουργείο και, να μπει, και μπαίνει έτσι μέσα στις υποθέσεις της κυβέρνησης. Φυσικά και θα πρέπει να επιμείνουμε ώστε να υπάρχουν οι κατάλληλοι πόροι σε επίπεδο των κοινοβουλίων μέσα στο πλαίσιο του ίδιου του εθνικού προπολογισμού, όπου οι δωρητές βεβαίως συμβάλλουν. Αυτέ είναι οι αρχικέ μου παρατηρήσεις, αλλά όπως σα είπα είναι μια εξαίρετη μελέτη που θα μας βοηθήσει στον προβληματισμό μας ε, για την αναθεώρηση του οδηγού ή στην πράσινο βιβλίο. Αν μου το επιτρέπετε, αν μπορεί να πάρει το λόγο και ο συνάδελφος από την ΕΚΟ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μάρκο Φορμεντίνη από την ΕΚΟ. Θα ήθελα να προσθέσω μερικά πράγματα βρίσκουμε ότι η έκθεση έχει ένα πλούσιο θα έλεγα και ενδιαφέρον σώμα και θα μας βοηθήσει και σε εμά στην εσωτερική μας εργασία. Θα λέγαμε ότι τα μεγάλα πνεύματα συναντώνται. Προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε μια ε, να κάνουμε μια αλλαγή σημαντική στον τρόπο ε, που λειτουργούμε όσον αφορά αυτή τη συζήτηση. Τρία σημεία θα θίξω. Πρώτον, υπάρχει, ο κύριος Κρεβέη το είχε πει, υπάρχουν παρεμβάσεις της Επιτροπής ε, για νομοθετική υποστήριξη σε πολλές χώρες το πρόβλημα το οποίο αναφέρεται και στην έκθεση είναι δύσκολο για την Επιτροπή να μονομερώσει ή με υποχρεωτικό τρόπο να, να προχωρήσει αυτό το θέμα το νομοθετικό βλέποντας και θέματα που έχουν να κάνουν με την ε, ανεξαρτησία σε σχέση με το ελεκτικό συνέδριο και με μηχανισμούς ελέγχου εξωτερικούς. Είναι αλήθεια ότι στις εσωτερικοί μας κατευθύνσεις γραμμές, ο ρόλος του Κοινοβουλίου, των Κοινοβουλίων δεν αναλύεται όσο θα έπρεπε. Αντιθέτως, και οι συνάδελφοι που είναι εδώ από πίσω, προσπαθούμε να προετοιμάσουμε κάποιες κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά την υποστήριξη κοινοβουλίων. και για το ρόλο όσον αφορά στις, ε, ε, τα θέματα που αφορούν τον προπολογισμό. Λοιπόν, υπάρχουν θέματα τα οποία θα προχωρήσουν γρήγορα τι επόμενους μήνες και θα ήταν σημαντικό όταν θα έχουμε θα συνεχίσει η συζήτηση για τη σύνταξη αυτή του ΙΣΙΚ έκθεσης, αγαστή συνεργασία με, το, με, το, με την Επιτροπή στα πλαίσια της Πράσινης Βίβλου, αλλά και σε συνεργασία και με άλλα μέσα που έχουμε στη διάθεση μας, να έχουμε ένα, θέλουμε να έχουμε ένα ε, ρεαλιστικό διάλογο με την Επιτροπή, να δούμε ποιες είναι οι κατευθυντήρες γραμμές της Επιτροπής πάνω σε αυτό το θέμα. Ευχαριστώ, ευχαριστώ η πρόεδρος. Κύριε Κόχ, έχετε το λόγο για να απαντήσετε. Thank uh, uh, Σας ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας. Ε, σε σχέση με την πρώτη ερώτηση, ερώτηση για τους όρους. Πρέπει να υπάρχουν όροι. Είναι μια, ε, μια θέση κλειδί όσον αφορά την διαχείριση κινδύνου. Το θέμα είναι κατά πόσο μπορούν να συμπεριληφθούν τα κοινοβούλια στους όρους αυτούς. Θα πρέπει να αξιολογήσουμε αναπερίπτωση την κατάσταση. Γιατί όπως είπα, το εκτελεστικό πρέπει να ελέγχει την πιθανή πλήρωση των όρων αυτών. Αν δούμε λοιπόν τους όρους, αν δούμε το, από το, υπό το φως της εξωτερικής, του εξωτερικού ελέγχου, θα πρέπει να υπάρχουν, γιατί κατά κάποιο τρόπο δίνει κανείς χρήματα σε μια κυβέρνηση. Αλλά θα πρέπει να δούμε αν αυτό εξισορροπείται από την εγχώρια, τον εγχώριο έλεγχο. Πράγμα που δεν συμβαίνει. Γι' αυτό και πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τον εγχώριο έλεγχο. Τι μπορούν να κάνουν οι δωρητές ώστε να μην μειωθεί ο εξωτερικός έλεγχος σε μακροπρόθεσμα. Και Δεύτερον, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας από τους μεγαλύτερους δωρητές και στηρίζει πολλούς προπολογισμού. Αν υπήρχε μια μείωση, νομίζω πως η Κομισιόν θα ήταν σε καλύτερη θέση να απαντήσει. Αλλά αυτό που είδαμε εμείς σε αυτές τις τρεις χώρες είναι ότι υπάρχει μικρή μείωση τον περασμένο χρόνο και δεν ξέρω αν αυτό έχει να κάνει με την ύφεση, αλλά μπορεί να το δει κανεί και σε άλλες χώρες ότι αντίθετα υπάρχει αύξηση. Ίσως η Κομισιόν λοιπόν να μπορούσε να απαντήσει την ερώτηση αυτή όσον αφορά την ενίσχυση των κοινοβουλίων. Θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε πως αυτή η μελέτη δεν είναι η σβάθο μελέτη της ενίσχυσης των κοινοβουλίων και γι' αυτό και στο παράρτημα έχουμε συμπεριλάβει το στις κατευθυντήριες γραμμές του OEDA στο Ηνωμένο Βασίλειο για το ποιες είναι οι κατευθυντήριες γραμμές για να δούμε ποια είναι πραγματικά η δυνατότητα ενίσχυσης των κοινοβουλίων. Έχουμε εξετάσει ωστόσο αυτές τις τρεις χώρες και αυτό που μπορούμε να πούμε σαφώς σε σχέση με τους πόρους και την έλλειψη δυνατοτήτων η εισαγωγή κοινοβουλευτικών γραφείων για τον προπολογισμό βοήθησε στο να αυξηθεί η δυνατότητα των κοινοβουλευτών να αναλύσουν και να ελέγξουν τον προπολογισμό. Όταν όμως μιλάμε για τα κοινοβούλια. Δεν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει ίδια, το ίδιο επίπεδο σε όλα τα κράτη. Ας πούμε στην Ασία το ίμιση των βουλευτών είναι αγράμματοι, αναλφάβητοι. Δεν μπορούμε να το συγκρίνουμε με την Κάνα, ας πούμε, που υπάρχει διαφορετικό επίπεδο κατανόησης. Αλλά θα πρέπει να υπάρξει στήριξη για αυτούς τους βουλευτές. Για παράδειγμα, στα γραφεία, τα κοινοβουλευτικά για τον προπολογισμό μπορούσαν να δώσουν αναλύσεις εκεί για τομεακέ τομεακά θέματα ας πούμε, για την παιδεία και σαφώς τα κοινοβούλια δεν μπορούν να τα καταφέρουν από μόνο τους. Δεν έχουν βοηθούς, δεν έχουν σχεδόν γραφεία. Είναι κάτι το οποίο θα μπορούσαν να βοηθήσουν οι δωρητές ώστε να ε, υπάρχουν καλύτερες συνθήκες. Οι δημόσιες ακροάσει επίσης είναι κρίσιμε. Θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι στην Γκάνα λειτουργεί καλά από ό,τι φαίνεται, γιατί η φήμη του Κοινοβουλίου βελτιώνεται. Ενώ στη Δομινικανή Δημοκρατία οι δημόσιε ακροάσει γίνονται, αλλά δεν λειτουργούν καλά, διότι τόσο άσχημη φήμη έχει το κοινοβούλιο που κανείς δεν ενδιαφέρεται. Αν θέλουμε πραγματικά να ενισχύσουμε λοιπόν θα πρέπει να δούμε ανακράτος τι συμβαίνει. Δεν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μία λύση για όλους. Επίσης ήθελα να πω σε σχέση με ένα άλλο ερώτημα ότι όταν εξετάσει κανείς την ενίσχυση των κοινοβουλίων και τα όσα άκουσα από την Κομισιόν τώρα νομίζω πως το να αυξηθεί η ισχύ των κοινοβουλίων μέσα στο πλαίσιο της στήριξη των προπολογισμών είναι πολύ σημαντικό. Ωστόσο, είναι παραπλανητικό το να σκέφτεται κανείς ότι οι κυβερνήσεις είναι διφθαρμένες ενώ το κοινοβούλιο όχι. Δηλαδή, δεν είναι ο ένα ο καλό και ο άλλο ο κακός. Θα πρέπει να προσθεθεί και ένα τρίτο στοιχείο που θα μπορούσε να είναι η φορείς, οι διάφοροι κοινωνικοί φορείς. Είναι σημαντικό να δούμε και αυτούς τους φορείς και να εξετάσουμε και τους μηχανισμούς των πολιτών όσον αφορά τον έλεγχο που κάνουν οι ίδιοι στα κοινοβουλιά τους. Πρέπει εδώ να γίνει περισσότερη δουλειά σίγουρα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Έχω ένα ανέκδοτο να σας πω, μια ιστορία όσον αφορά τον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Βρισκόμουν σε ένα νησί που δεν θέλω να σας αναφέρω με 125.000 κατοίκους όλους και όλους και έδινα ένα μάθημα στο κοινοβούλιο για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Μόλις να βρει πετρέλαιο εκεί και θεωρήσαμε πως ήταν πολύ σημαντικό να ευαισθητοποιηθεί το Κοινοβούλιο στην, για τη σημασία των συμβάσεων που πρόκειται να συναυθούν. Στο τέλος της ομιλίας μου, της ηγησής μου, είχα δύο ερωτήσεις. Η πρώτη ήταν, κυρία Ζολή, πιστεύετε πραγματικά ότι θα είμαστε, οι, ότι, ότι θα είμαστε οι πρώτοι που δεν θα πλουτίσουμε και έπειτα... Ποια είναι τα όρια για την δήλωση εισοδημάτων. Για να σας πω μόνο ότι ο δρόμος που πρέπει κανείς να διανύσει για να φτιάξει κοινοβουλευτικό έλεγχο είναι πολύ πολύ μακρύς και ότι δεν θα πρέπει να παραμελούμε και την ε, δημιουργία και να δουλέψουμε και για τα ελεγκτικά συνέδρια και τον έλεγχο από εμά, εμάς τους ίδιους. Και ότι αυτός ο δρόμος του κοινοβουλευτικού ελέγχου θα μας πάρει δεκαετίες Ας στραφούμε τώρα στο άνατο σημείο της ημερήσιας διάταξης που είναι τα πρακτικά της αντιπροσωπείας μας, της κοινή αντιπροσωπείας μεταξύ της Επιτροπής μας, ε, της Επιτροπής Προπολογισμού και της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων στην Παλαιστίνη και στο Ισραήλ από τις 24 έως τις 28 Μαΐου φέτος. Θα θυμάστε ότι η επίθεση ε, εναντίον του στο Λίσκο έγινε τη νύχτα της 30ης προς την 31η Μαΐου και αυτό έδωσε ιδιαίτερες αποχρώσεις και σημασία στο δικό μας ταξίδι. Στόχος της αντιπροσωπείας μας, της κοινής αντιπροσωπείας, ήταν να αξιολογήσουμε επιτόπου την πολιτική και ανθρωπιστική κατάσταση και να προσπαθήσουμε να εκτιμήσουμε τον αντίκτυπο της δικής μας οικονομικής συμβολής γιατί όπως το γνωρίζουμε όλοι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο μεγαλύτερος δωρητής εν γέννη για την υπεριορδανία ε, και την Γάζα και συμβάλλουμε με πάνω από 500 εκατομμύρια ευρώ. Υπάρχει μια έκθεση για αυτή την αποστολή που έχει προετοιμαστεί και έχει διανεμηθεί. Προτείνω λοιπόν να σας κάνω μια σύντομη ε, προφορική αναφορά και έπειτα να σας δώσω το λόγο για τις παρατηρήσεις σας και τις ενδεχόμενες ερωτήσεις σας. Συμφωνείτε να σας μιλήσω για πέντε λεπτά για να σας πω τα όσα συνέβησαν. Μάλιστα. Il était d'abord important de constater en Cisjordanie qu'ils ont connu en 2009 une croissance importante. Το 2009, όπως ε, στην Παλαιστίνη, παρατηρήθηκε μία αύξηση σημαντική του ΑΕΠ και αυτό οφείλεται στην χαλάρωση των Ισραηλινών περιορισμών, αλλά επίσης στην προσπάθεια των Παλαιστινιακών Αρχών όσον αφορά την διακυβέρνηση, την ασφάλεια, την καταπολέμηση της διαφθοράς και το κράτος δικαίου. αν θέλουν να διατηρήσουν αυτό το εξαιρετικό ποσοστό ανάπτυξης, αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να ε, υπάρχει πρόσβαση στη ζώνη σε για τον επόμενο χρόνο και βεβαίως θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να ανοίξει με ποσοστώσεις ε, τα την αγορά της στα παλαιστινιακά προϊόντα. Ε, κάτι τέτοιο θα ήταν πολύ ευπρόσδεκτο. Βεβαίως ε, είχαμε επαφές με τον Πρωθυπουργό Φαγιάντα και μας είπε ότι θα μπορούσε να μπορέσει να λειτουργήσει το Παλαιστινιακό κράτος ε, κανονικά από το 2011 και ότι αυτό θα είχε συνέπειες όσον αφορά τον στήριξη στον προπολογισμό που δίνουμε στην Παλαιστινιακή Αρχή. Πράγματι, αυτή η στήριξη είναι η μεγαλύτερη κατακεφαλήν στον κόσμο. θα επιθυμούσε, αν το Παλαιστινιακό Κράτος λειτουργήσει το 2011, να προσανατολίσουμε ένα μεγάλο τμήμα τη στήριξή μα στην ε, στήριξη προγραμμάτων του ιδιωτικού τομέα, ώστε η οικονομία να μπορέσει να λειτουργήσει και να οδηγήσει στην πληρωμή των υπαλλήλων από την ίδια την Παλαιστινική Αρχή. Πολύ σαφή συμβούληση, λοιπόν ότι να προσανατολιστεί η ενίσχυσή μας στον ιδιωτικό τομέα. Είναι βέβαιο πως η συνεργασία με το Ισραήλ είναι πολύ σημαντική για να μπορέσει η Παλαιστινιακή Αρχή να φτιάξει τις κατάλληλες δομές, αλλά είναι σαφές πως αυτό δεν μπορεί να υποκαταστήσει τις ειρηνευτικές ε, διαπραγματεύσεις που θα πρέπει να καταλήξουν στην δημιουργία δύο κρατών. και η προσέγγιση που στηρίζει ο Πρωθυπουργό στο bottom-up δεν είναι βιώσιμη παρά μόνο αν βγούμε αν τελειώσει η κατοχή. Θα πρέπει να πω πως εντυπωσιαστήκαμε από την βία που επικρατεί στο τοπίο, από την βία των τυχών που χωρίζουν την Ανατολική Ιερουσαλήμ από την Δυτική Όχθη και επίσης γιατί βλέπουμε στο... είδαμε το κλείσιμο των ε, δρόμων. Δημιουργούν δηλαδή χωριστούς δρόμους για τους Παλαιστινίους, οι οποίοι ε, κλείνονται από, ε, από φράγματα από τις δύο πλευρές. Δηλαδή η, γλώσσα του τοπίου λέει ότι κατασκευάζεται ένα κράτος apartheid. Έπειτα, εννέα από την αντιπροσωπεία μας πήγαν στην Γάζα. Θα θυμάστε πως δεν είχαμε την Ισραηλινή άδεια για να μπούμε στην λωρίδα της Γάζας από την Ισραηλινή πλευρά, άρα υποχρεωθήκαμε να πάμε από το Κάιρο και να περάσουμε από το ε, Ράφα συνάντηση, ή μάλλον η επαφή με τη Γάζα ήταν ένα σοκ. Δεν υπάρχει άλλο, άλλη λέξη για να περιγράψει κανείς το τι συμβαίνει εκεί. Υπάρχουν ξεκάθαρα ίχνη του αποκλεισμού, των βομβαρδισμών. Το 80% των σχολείων δεν έχουν μπορέσει να νοικοδομηθούν. Και όλη την ώρα βομβαρδίζονται οι υπόνομοι, πράγμα που που οδηγεί στο ότι οι υπόνομοι οδηγούν κατευθείαν στη θάλασσα, πράγμα το οποίο είναι υγειονομικό κίνδυνο και διαπιστώσαμε πόσο ανθεί... Είναι το, η κατασκευή σειράγγων Υπάρχουν πάρα πολλέ σειράγγε στην Γάζα και μπορεί κανείς να βρει τα πάντα. Υπάρχει μια έντονη αντίθεση μεταξύ των σχεδίων ανοικοδόμησης που είδαμε υπό την αιγίδα του ΟΗΕ που κατασκευάζει καταλήματα για 12 Παλαιστινίους και που έχει σταματήσει, έχει ανασταλεί αυτή η κατασκευή γιατί δεν έχουν τσιμέντο για να μπορέσουν να κατασκευάσουν αυτά τα καταλήματα τη στιγμή που αυτά τα καταλήματα χρηματοδοτούνται πλήρως από τους ε, δωρητές και πολλά από αυτά τα κτίρια για τα καταλήματα ήταν πολύ κοντά στο να συμπληρωθούν. Ο ΙΕ αρνήθηκε να πάρει τσιμέντο από την μαύρη αγορά, ενώ συγχρόνως βλέπουμε η Χαμάς να κατασκευάζει κτίρια, χρησιμοποιώντας προφανώς την μαύρη αγορά. Συναντηθήκαμε επίσης και με εκπροσώπους της ε, Τράπεζας της Παλαιστίνης στη Γάζα, που μας είπαν ότι δεν υπάρχει ουσιαστικά τραπεζική δραστηριότητα στη Γάζα δεν υπάρχει επιχειρηματική ζωή στη Γάζα. Είδαμε ότι η τράπεζα παρόλα αυτά αποκόμιζε κέρδη από τις δραστηριότητές της στην Δυτική Όχθη αλλά όχι στη Γάζα. Γιατί στη Γάζα δεν μπορεί να υπάρξει εμπόριο και φυσικά δεν μπορεί να υπάρξει και τραπεζική δραστηριότητα. Είναι ένα ακόμα γεγονός το οποίο προέρχεται από, την, από τον αποκλεισμό της Γάζας. Η Κομισιόν έχει υπολογίσει τι κοστίζει αυτός ο αποκλεισμός της Γάζας για τη λόγια της Γάζας. Οι υπολογισμοί είναι ότι ο αντίκτυπος αυτού του αποκλεισμού είναι περίπου 514 δισεκατομμύρια ευρώ και περίπου 12 εκατομμύρια για τα σχέδια υποδομών αυτό είναι μια απώλεια συνολική για όλο τον κόσμο. Εμείς κάναμε πολύ σημαντικές συναντήσεις με την Ούνρα, τον φορέα για την ανακούφιση των προσφύγων και είδαμε ποια είναι η κατάσταση των σχολείων. Η, η Ούνρα είναι, αυτή, η ο που εξασφαλίζει την σχολική εκπαίδευση στο δημοτικό όλων των παιδιών στη Γάζα. Αυξάνει κάθε χρόνο ο αριθμό των παιδιών που πηγαίνουν στο σχολείο, γιατί 50% του πληθυσμού στη Γάζα έχει ηλικία κάτω από 18 ετών, επομένω είναι σε σχολική ηλικία. Υπάρχουν δεκάδε χιλιάδων νέων μαθητών κάθε χρόνο, αλλά δεν μπορούν να οικοδομήσουν νέε αίθουσε γιατί δεν έχουν ε, οικοδομικά υλικά και δεν μπορούν καν με σταθερό προπολογισμό να δημιουργήσουν νέες νέες τάξεις με το να λειτουργούν οι τάξεις 24 ώρες 24 γιατί δεν έχουν λεφτά να πληρώσουν τους καθηγητές. Είναι λοιπόν μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω του αποκλεισμού, αλλά επίσης και λόγω της απώλειας της ε, αξίας του ευρώ έναντι του δολαρίου. Βρισκόμαστε λοιπόν σε μια επισφαλή κατάσταση από οικονομική απόψη και χρειάζονται νέες χρηματοδοτήσεις. το γεγονό ότι δεν υπάρχει εδαφική συνέχεια με τη Δυτική Όχθη και αυτό αποτελεί ένα μεγάλο πρόβλημα μέσα στην προοπτική της επανένωσης του Παλαιστινιακού κράτους που θα περιλαμβάνει και τη Γάζα και την Δυτική Όχθη και θα πρέπει στο μέλλον να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρξει αυτός ο διάδρομος μεταξύ των δύο τμήματων όπως προβλεπόταν και από τη Συμφωνία του 2005. Η αντιπροσωπεία μας την Παρασκευή πρωί όταν φύγαμε πριν φύγουμε μάλλον, κάναμε μια ανακοίνωση τύπου. Δεν είχε γίνει ακόμα η επίθεση κατά του ανθρωπιστικού στολίσκου και με ομοφωνία, όχι μόνο αυτών που ήταν παρόντες στη Γάζα, αλλά και αυτών που είχαν παραμείνει στην Ιερουσαλήμ, ζητήσαμε να υπάρξει τέλος του αποκλεισμού, να υπάρξει άμεσο πέρας του αποκλεισμού της Γάζας. Βέβαια, η συνέχεια των γεγονότων κατέδειξε πόσο σημαντικό είναι από πολιτική άποψη να γίνει πραγματικότητα αυτή η άρση του αποκλεισμού. Επίσης, η ανακοίνωσή μας στον τύπο ζητούσε από την Ευρώπη να προχωρήσει μια πολιτική δράση. Ομόφωνα, η αντιπροσωπεία μας διαπίστωσε ότι θα πρέπει να έχουμε ένα κοινό ψήφισμα το οποίο να έχουμε τη βάση μάλλον το ψήφισμα το οποίο ψηφίστηκε την προηγούμενη Πέμπτη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το οποίο ζητούσε την άρση του αποκλεισμού της Λωρίδας της Γάζας. Με συμφωνία των επιτροπών οι οποίοι ενεπλέκονται σε αυτή την αποστολή. Νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό να λάβει χώρα και στο μέλλον. Θα πρέπει να διατηρήσουμε αυτή την ενότητα δράσης μεταξύ μας. Προσκαλέσαμε τον Τζον Κιν ο οποίος είναι ο υπεύθυνο της Ούνρα, να έρθει να μας μιλήσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό θα γίνει σε συνεργασία και με τις δύο άλλες επιτροπές. Στις 5 Ιουλίου θα λάβει χώρα αυτή η συνάντηση. Και θα έχουμε και τον Πρωθυπουργό Φαγιάτ, ο οποίος θα μιλήσει ενώπιον αυτών των επιτροπών στις 13 Ιουλίου. Σας παρακαλώ λοιπόν να καταγράψετε αυτά τα, αυτές τις δύο συναντήσεις γιατί αυτή είναι η πρώτη εκδήλωση της κοινή θέληση των τριών επιτροπών. Θέλω να τονίσω λιγάκι τον πολιτικό ρόλο που πρέπει να έχουμε για να υπάρξει μια δραστηριοποίηση και δυναμικοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαστε ο μεγαλύτερος χορηγός προς την Παλαιστινιακή Αρχή. Είμαστε επίσης και ο πρώτος εμπορικός εταίρος του Ισραήλ. Και εδώ υπάρχει μια βία αντίφαση μεταξύ αυτής της κατάστασης και της πολιτικής απουσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ειρηνευτική διαδικασία. Εξακολουθεί ακόμα και σήμερα να είναι ακατανόητο αυτό. Γι' αυτό μας φαίνεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα πρέπει να φοβηθεί να προσφύγει σε μία εξάρτηση έναντι των τοπικών φορέων και έναντι του κουαρτέτου επίσης. Ζητούμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να λάβει τις απαραίτητες διπλωματικές πρωτοβουλίες και είπα σήμερα το πρωί ότι υπάρχει ήδη μια απαρχή της άρσης του αποκλεισμού και αυτό είναι αποτέλεσμα των διπλωματικών δράσεων που έφερε σε πέραση η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και άλλοι εταίροι. Θα πρέπει εμείς όμως να φροντίσουμε η άρση του αποκλεισμού να είναι πλήρης και να υπάρχει ελεύθερη διέλευση για τα εμπορεύματα, να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε τον τωρινό κατάλογο προϊόντων όπου αυτά τα οποία δεν επιτρέπονται εκπεφρασμένα απαγορεύονται όπως σήμερα, να έχουμε μόνο ένα κατάλογο απαγορευμένων ειδών. Θα πρέπει επίσης να επανεξετάσουμε την παρουσία μας μέσα στο κουαρτέτο για να υπάρξει και αναθεώρηση της εντολής του κουαρτέτου και να αναθεωρήσουμε καλύτερα το ρόλο και τα αποτελέσματα που επέτυχαν οι εκπρόσωποι του κουαρτέτου διότι ένα τμήμα της αποστολής του εκπροσώπου του κουαρτέτου χρηματοδοτείται από εμάς. Και μετά από τα συμπεράσματα του Συμβουλίου του 2009 θα πρέπει να προτείνουμε μια στρατηγική για την Ιερουσαλήμ για να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής των πολιτών, των κατοίκων της και να εξασφαλίσουμε και τη συνέχιση της παρουσίας των χριστιανών και μουσουλμάνων κατοίκων στο ανατολικό τμήμα της Ιερουσαλήμ με προγράμματα τα οποία αντιμετωπίζουν την ανάγκη των νέων, την εκπαίδευσή τους, την πολιτιστική λειτουργία και την τοπική διακυβέρνηση. Με την ευκαιρία λοιπόν αυτή θα πρέπει να διατυπώσουμε μια πολιτική πιο φιλόδοξη και πιο συνεκτική γιατί τώρα η ύπατη εκπρόσωπος μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα πιο αποτελεσματικό διπλωματικό εργαλείο. Έχει αυτή τη στιγμή υπό την εποπτεία της την οικονομική βοήθεια και όλα τα εργαλεία της ΚΕΠΑ. Έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει και τον ειδικό απεσταλμένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή αυτή. Εν κατακλείδη πιστεύω ότι πολύ σπάνια μια αποστολή αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ήταν τόσο πλούσια σε διδάγματα και πολύ σπάνια στο παρελθόν είχαμε τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε μια τόσο στεναρή συμφωνία και συνεννόηση μεταξύ των διαφόρων επιτροπών και των διαφόρων πολιτικών ομάδων. Θεωρώ λοιπόν ότι ήταν μια πάρα πολύ επιτυχής αποστολή και πολύ σημαντική. Και σας προτείνω να συνεχίζετε τις προσπάθειές σας ώστε να εξασφαλίσουμε ότι η ύπατη εκπρόσωπος καθώς και η Κομισιόν θα ακολουθήσουν και θα ενστερνιστούν τις ε, συστάσεις που περιλαμβάνει το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ. Έχουμε μια ομάδα επισκεπτών. Μόλι μου είπαν ότι η ομάδα των επισκεπτών που μπήκαν εδώ στην αίθουσα είναι δημοσιογράφοι από τη Σρι Λάνκα. Σας καλωσορίζω λοιπόν θερμά για να παρακολουθήσετε το πέρας της σημερινής μας συνεδρίασης. Κύριε Κάσμαν, είχατε ζητήσει το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω ότι η επίσκεψη αυτή δεν θα μπορούσε να είναι πιο επίκαιρη. Διαβάζοντας την έκθεση που προετοιμάσατε θα πρέπει να πω πως είναι κάπως απογοητευτικό, καταθλιπτικό. Φαίνεται να βλέπουμε δύο κράτη που και τα δύο είναι, αισθάνονται ότι είναι υποεπίθεση. Ο ένας ε, αποφάσισε να αντιδράσει επιθετικά, ενώ ο άλλος παθητικά. Και νομίζω πως ε, είναι παράξενη αυτή η κατάσταση και δεν υπάρχει καθόλου ισορροπία και δεν καταλαβαίνω γιατί έχει γίνει αυτό. Είναι πολύ ανησυχητικό και όντως ε, τα όσα ε, μαρτυρίες γράφεται εδώ στην έκθεση για αυτές τις ΜΚΟ που πρέπει να δηλώνουν οποιοδήποτε πόρο πηγή δημόσιας χρηματοδότησης ας πούμε και αν τα χρήματα προέρχονται από ιδιώτες που πολλές από τις, τις τους επικισμούς δέχονται, δεν πρέπει να δηλώνονται. Φαίνεται δηλαδή να υπάρχει μια λογοκρισία και αποκλεισμό των ΜΚΟ από τη σωστή εκπροσώπηση της κοινωνίας των πολιτών. Και επίσης βρίσκω πολύ ενδιαφέρουσα τη συζήτηση που έγινε ε, για το θέμα του κατά πόσο το Ισραήλ είναι εβραϊκό κράτος ή κράτος το οποίο είναι πολυεθνικό. Και τα συμπεράσματα εκεί φαίνεται να αντικατοπτρίζουν ότι υπάρχει διχόνοια εντό τη Κνέσετ όσον αφορά αυτή την προσέγγιση. Επίσης είναι εντυπωσιακό ότι τα μέλη της Κνέσετ ανέφεραν την άποψη ότι οι αυξανόμενοι και συνεχιζόμενοι επικισμοί δεν αποτελούν απειλή για οποιαδήποτε συμφωνία. Φαίνεται δηλαδή ο κόσμος να ζει σε ένα παράλληλο σύμπαν, όπου οι διάφορες ενέργειες αναμένατε ότι δεν θα έχουν ε, αντίδραση, θα μείνουν αναπάντητες. Ε, ε, πολύ ενδιαφέρουσα λοιπόν η έκθεσή σας και θα ήθελα να ακούσω αν εσείς αισθανθήκατε καθώς ήσασταν εκεί αν η πολιτική συζήτηση επηρεάστηκε από το περιστατικό της, του, του, Στολίσκου, ανάμεσα δηλαδή στην, αν υπήρξε σχετικέ συζητήσει ανάμεσα στην Ιουδαϊκή κοινότητα, την ΚΝΕΣΕΔ και αν υπάρχει βάσιμη πιθανότητα για επίλυση του προβλήματος ανάμεσα στις δύο πλευρές, αν αναμένει κανείς δηλαδή ότι η Παλαιστινιακή πλευρά θα, θα, θα παρουσιαστεί ως μια γενομένη. Να ακούσω επίσης παραπάνω πράγματα. Ε, ε, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω τη λέξη αυτή, αλλά αυτή την ανάπτυξη του καθεστώτος Απαρχάιντ, όπου φαίνεται να υπάρχουν ε, διαχωριστικά τείχη ανάμεσα στους μεν και στους δε. Αν δεν χρησιμοποιήσουμε την επιρροή μας ώστε να γίνουν αλλαγές, όπως κάναμε την περασμένη εβδομάδα, να είμαστε δηλαδή τμήμα μιας διεθνούς έκκλησης για αλλαγή, τότε πραγματικά σπαταλάμε τις επενδύσεις που κάνουμε στην Παλαιστίνη και στο Ισραήλ. Σας ευχαριστώ για την εξαιρετική σας έκθεση ωστόσο και ε, για το ότι μας ενημερώσατε. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε για την εκθεσή σας. Ήταν εντυπωσιακό αυτό που είπατε, αλλά συγχρόνως ήταν και καταθλιπτικό. <clears throat> Γιατί κάνει σαφές ότι το Ισραήλ δεν πρόκειται να αλλάξει προς τα βελτίο την ε, στάση του, αλλά φαίνεται ότι θα επιμείνει στην πολιτική επικισμών. Αυτό είναι ένα σαφές επιθετικό στοιχείο της πολιτικής του Ισραήλ. Το πρόβλημα δεν είναι τόσο πολύ το πρόβλημα της Λόριδας της Γάζας, όσο η πρόθεση των επικισμών στη Δυτική Όχθη από την πλευρά του Ισραήλ και εδώ φαίνεται ότι είναι απόλυτα αδύναμη και αβοήθητη η Ευρωπαϊκή Ένωση και το κουαρτέτο. Χθες δεν μπόρεσε να πάει ο Γερμανός Υπουργός Ανάπτυξης στην Γάζα για να παρακολουθήσει, για να επισκεφθεί ένα γερμανικό σχέδιο ε, ανάπτυξης. Δεν πρόκειται για ένα άτομο το οποίο είναι εναντίον του Ισραήλ είναι αντιπρόεδρος του Ιδρύματος Φιλίας μεταξύ Ισραήλ και Γερμανίας και παρόλα αυτά είχε να αντιμετωπίσει την στάση αυτή του Ισραήλ που δείχνει πόσο απομονωμένο είναι πια το Ισραήλ. Θα πρέπει να σκεφτούμε πώς θα δράσουμε εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι ένα σημαντικό στοιχείο, με ένα σημαντικό δείγμα της θέλησής μας είναι να προσκαλέσουμε Παλαιστίνιους να έρθουν εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μια άλλη δυνατότητα είναι να ανακοινώσουμε περαιτέρω επισκέψεων επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Δυτική Όχθη και στη Γάζα. Όπως είπαμε, είναι μια πάρα πολύ καταθλιπτική κατάσταση που περιγράφεται από την έκθεση και προς το παρόν εγώ δεν μπορώ να δω καμία δυνατότητα εξόδου από αυτή την κατάσταση διεξόδου. Ευχαριστώ. Κύριος Βάγγελ. Ευχαριστώ. Όταν θέλω να πω κάτι το οποίο έχει συγκινησιακό χαρακτήρα, εγώ πρέπει να επιστρέφω στη μητρική μου γλώσσα. Νομίζω ότι αυτή η έκθεση της κυρίας Ζολή είναι θαυμάσια. Αντανακλά με πλήρη τρόπο την ε, πολύ καλά προετοιμασμένη επίσκεψη που έκανε η αντιπροσωπεία μας. Οι συνομιλητές μας έτυχαν μιας προσεκτικής επιλογής και επειδή και εγώ ήμουν μέλος αυτής της αντιπροσωπείας και μάλιστα του τμήματος που πήγε στη Γάζα, θα πρέπει να τονίσω τα εξή στοιχεία. Στην Παλαιστίνη, στο Ισραήλ, στη Λωρίδα της Γάζας, σε όλα αυτά τα εδάφη υπάρχουν εξαίρετοι εκπρόσωποι της διεθνούς κοινότητας που μας έδωσαν πολλά στοιχεία και πολλές πληροφορίες για την πραγματική κατάσταση που επικρατεί επί επιτοπίως. Ιδίως αναφέρομαι στους ε, εκπροσώπους της ΟΣΑ και της, ε, των Ηνωμένων Εθνών. Η παρουσία τους λοιπόν είναι πάρα πολύ επωφέλης και τη θυμάμαι πάντα μετά από αυτή την αποστολή. Κύριε Πρόεδρε, δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο μαζί σας όταν τονίζετε ότι ήταν πάρα πολύ επίκαιρη η επίσκεψη αυτή. Γιατί κατά κάποιο τρόπο εμείς γίναμε κομμάτι των δραματικών γεγονότων που έλαβαν χώρα στα Παλαιστινιακά εδάφη. Συγχρόνως όμως πιστεύω ότι επιτύχαμε να επηρεάσουμε τα τεκτενόμενα μετά από αυτήν την τόσο ατυχή επίθεση στον ανθρωπιστικό στόλο που πήγαινε προς τη Λωρίδα της Γάζας. Σήμερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στα μέσα ενημέρωσης και μέσα στη διεθνή κοινότητα, χάρη σε αυτή την επίσκεψη μπορούμε να συζητήσουμε με πιο αξιόπιστο τρόπο τις σχέσεις μεταξύ του Ισραήλ και του Παλαιστινιακού λαού. Ο συναδελφός μου, κ. Κάσμαν, έθεσε ένα ερώτημα το οποίο για μένα είναι παραπάνω από δικαιολογημένο. Πράγματι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη διατύπωση του apartheid, γιατί πολλοί από εμά οι οποίοι συμμετάσχαμε σε αυτή την αποστολή σκεφτόμασταν ακριβώς αυτή τη χρήση. Εγώ έχω χρησιμοποιήσει πολλές φορές τα άρθρα μου το, τη διατύπωση apartheid. Δεν είναι apartheid το να έχουμε κάποιους οι οποίοι πιστεύουν ότι η ζωή τους στα εδάφη τα Παλαιστινιακά μπορεί να βασιστεί σε ένα διαχωρισμό με τύχη, με παράλληλους δρόμους, με παράλληλα πεζοδρόμια, με παράλληλα, ε, παράλληλους παιδικούς σταθμούς και χώρους παιχνιδιών για τα παιδιά. Όλα αυτά δημιουργούν και εκτρέφουν μία απομάκρυνση, μία ένα διαχωρισμό από τους συνανθρώπους τους. Αυτοί οι οποίοι θα πρέπει να συνεπάρχουν και να συμβιούν δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα. Το ζωή πρέπει να κατανοήσει κάποτε ότι δεν μπορεί με τύχη να απομονώσει τον εαυτό του από τους γείτονές του και ούτε μπορεί να το κάνει χρησιμοποιώντας μια πολιτική διακρίσεων κατά των Παλαιστινίων. Αυτά τα λέω όχι γιατί είμαι εχθρικός ή επικριτικός κατά του Ισραήλ. Μερικές φορές μπορεί να το θεωρούν οι διπλωμάτες του Ισραήλ ή κάποιοι από τους συναδέλφους μου εδώ στο Κοινοβούλιο. Εγώ ανησυχώ για ένα άλλο λόγο. Εγώ ανησυχώ γιατί χωρίς μια σύγχρονη προσέγγιση και χωρίς μια διαφορετική κατανόηση αυτού του πολύπλοκου θέματος δεν θα μπορέσει να υπάρξει ποτέ ειρήνη ούτε στη Μέση Ανατολή ούτε σε άλλα μέρη του κόσμου όπου η, το αδιέξοδο στις σχέσεις Ισραήλ και Παλαιστινίων δημιουργεί νέες αντιπαραθέσεις ακόμα και επιθέσεις τρομοκρατικού χαρακτήρα και τέτοιου είδους φαινόμενα. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτή η επίσκεψη της αντιπροσωπείας μας, της αντιπροσωπείας των τριών επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ήταν πάρα πολύ επίκαιρη και συμφωνώ με την Πρόεδρό μας ότι έχουμε εξασφαλίσει την πλήρη σύμνοια μεταξύ των τμήματων της αντιπροσωπείας, πέρα από πολιτικές ομάδες, πέρα από συμμετοχή σε μια συγκεκριμένη επιτροπή. Και νομίζω ότι αυτός είναι ο σωστός τρόπος για το Κοινοβούλιο μας και για την Ευρωπαϊκή Ένωση να προχωρήσει και να δώσει προστιθέμενη αξία σε όλες τις προσπάθειες οι οποίες έχουν σαν στόχο να ξεπεράσουν το αδιέξοδο της Μέσης Ανατολής. Η πολιτική που ακολουθεί ο Πρωθυπουργός κ. Φαγιάτ μας δίνει την ελπίδα ότι ίσως θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα νέα στοιχεία. Ένα από αυτά τα νέα στοιχεία είναι η ανάγκη να υπάρξει ένα Παλαιστινιακό κράτος. Μέσα σε μια ατμόσφαιρα μυσαλλοδοξίας και αντιπαράθεσης, η πολιτική του κ. Φαγιάτ μπορεί να οδηγήσει σε μια βελτίωση. Διάβασα σήμερα το πρωί ένα άρθρο από τον πρώην Γενικό Γραμματέα του Ισραηλινού Υπουργείου Άμυνας, ο οποίος χαιρετίζει την ιδέα αυτή του να υπάρξει ένα, ένα ανεξάρτητο κράτος Παλαιστινίων. Είπε ότι αυτό κινδυνεύει να επικριθεί ιδιαίτερα στη χώρα του, αλλά λέει ότι μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούμε εμείς να δημιουργήσουμε ένα πραγματικό και ισοδίκαιο διάλογο μεταξύ του κράτους του Ισραήλ και των Παλαιστινίων. Να υπάρχουν δύο κράτη, δύο πραγματικότητες, δύο οντότητες ένας διάλογος ο οποίος θα είναι αντίστοιχος με το διάλογο μεταξύ Ισραήλ και Συρίας, δηλαδή μεταξύ δύο γειτόνων και όχι ένας διάλογος ο οποίος βασίζεται σε εσωτερικά θέματα μονάχα. Υπάρχει λοιπόν αυτό το δίλημα και νομίζω ότι η επίσκεψή μας μας επέτρεψε να έχουμε μια καλύτερη επίγνωση της επιτόπιας κατάστασης. Εγώ προσωπικά πρέπει να πω ότι απογοητεύτηκα πάρα πολύ με τον διάλογο που έλαβε χώρα στην Κνέσετ. Μόνο δύο μέλη της Ισραηλινής Βουλής θεώρησαν ότι ήταν χρήσιμο να συναντηθούν μαζί μας και είναι φυσικά και οι δύο μέλη κομμάτων της αντιπολίτευσης. Μέσα σε αυτό το σύντομο διάλογο που είχαμε μεταξύ τους, μαζί τους, διαπιστώσαμε αυτό το οποίο διαπιστώσατε και εσείς ήδη, ότι υπάρχει ένα οξύδηλημα για το κατά πόσο το Ισραήλ θα πρέπει να είναι ένα εβραϊκό κράτος ή ένα κράτος που περιλαμβάνει όλους τους πολίτες του Ισραήλ. Το Σλοβενικό Σύνταγμα λέει ότι η Σλοβενία είναι το κράτος των Σλοβαίνων, αλλά έχουμε ένα ποσοστό 20% του πληθυσμού μας που αποτελείται από διάφορες μειονότητες. Αυτό ήθελα να τονίσω, αυτό προσπάθησα να τονίσω και εναντίον των Ισραηλινών συνομιλητών μα. Μακρηγόρησα πολύ, κυρία Πρόεδρε, και θα ήθελα κατακλείδη να πω το εξή. Σε ό,τι αφορά τα πολιτικά αυτά διλήμματα, κάτι πάντα με εντυπωσίαζε ιδιαίτερα. Όταν μιλάμε με τους εκπροσώπους, τους εκλεγμένους εκπροσώπους του Παλαιστινιακού λαού στη Ραμάλα, εμείς τους ρωτήσαμε πώς θα μπορούσε να επέλθει αυτή η εσωτερική συμφιλίωση μεταξύ των Παλαιστινιακών φατριών. Είπανε πολύ εύκολα. Μπορούμε να επιτύχουμε την συμφιλίωση. Μπορούμε να ξεκινήσουμε και μια νέα εκλογική διαδικασία. Θα αναγνωρίσει όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση τα αποτελέσματα αυτής της νέας εκλογικής διαδικασίας. Αυτό είναι το κέριο θέμα. Εμείς δεν μπορούμε να αρνηθούμε στο λαό της Παλαιστίνης το δικαίωμα που έχει οποιοδήποτε έθνος στον κόσμο να εκλέξει δημοκρατικά τους εκπροσώπους τους με μια δημοκρατική εκλογική διαδικασία. Αν εμείς δεν είμαστε πεπισμένοι ότι οι Παλαιστίνοι έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν μόνοι τους τους εκπροσώπους τους, όπως μπορούν να το κάνουν εξάλλου και οι Ισραηλινοί, είτε μας αρέσουν οι εκπρόσωποι τους ή όχι, αν δεν αναγνωρίσουμε αυτό το γεγονός, δεν θα μπορέσουμε ποτέ να καταλήξουμε σε μια λύση. Ευχαριστώ πολύ. Um, Ο Γκέι Μίτσελ. Εγώ θα προσπαθήσω να περιοριστώ στα σχόλιά μου στην ανθρωπιστική κατάσταση. Όσο αυστηρά λόγια έχω να πω για τους Ισραηλινούς, θέλω να τα πω κατηδίαν. Γιατί αν κανείς χρησιμοποιεί ε, αλλά εξ αποστάσεως δεν κάνει και μεγάλη διαφορά. Ακόμα και αν έχουμε τις μεγαλύτερες, καλύτερες προθέσεις στον κόσμο, οι οδηγίες που τους δίνουμε δεν λειτουργούν. Είπε κάποιο, ε, εγώ μπήκα σε ένα πολιτικό κόμμα στις, ε, όταν ήμουν ακόμα έφηβος λόγω των προβλημάτων που είχαμε στην Ιρλανδία αν πάει κανείς σε μέρη του Μπελφάστα θα δείτε ότι ανάμεσα στο Σάνκιλ και την, ε, την άλλο δρόμο που αν το δει κανείς από το Δουβλίνο ή από την πλευρά το, ε, σε, δημοκρατία της Ιρλανδίας ε, βλέπει μεγάλη διαφορά. Μας πήρε 30 χρόνια ανάμεσα στη συμφωνία της ε, Μεγάλης Παρασκευής και τη συμφωνία του Μπέλφας να καταφέρουμε στα όσα είχαμε συμφωνήσει το 1973. Ό,τι και τα πούμε, ό,τι και το ονομάσει κανείς, όλοι γνώριζαν ποια θα ήταν η λύση. Και εδώ όλοι γνωρίζουν ποια θα είναι η λύση, ότι θα είναι μια λύση δύο κρατών και ότι αυτό πρέπει να είναι το αποτέλεσμα. Τώρα σε σχέση με τα όσα υπόθηκαν, από, την, από ό,τι κατάλαβα, το ανώτατο δικαστήριο του Ισραήλ είναι πολύ ανεξάρτητο, δεν, δεν ακολουθεί τις ε, κυβερνητικές γραμμές, αλλά αν δει κανείς την λύση των δύο κρατών θα δείτε ότι θα έχει ε, ένα εβραϊκό υπόβαθρο, δεν είναι όλοι οι Εβραίοι εξάλλου θρησκευόμενοι και θα υπάρχει μια, ένα άλλο κράτος που θα είναι αραβικό και χριστιανικό. Θα υπάρχει δηλαδή, εν πάση περιπτώσει, αραβική κουλτούρα. Τα ίδια θέματα λοιπόν που προκύπτουν για το εβραϊκό κράτο θα πρέπει να θυγούν και για το αραβικό κράτος σε το χρόνο βεβαίως. Εγώ καλωσορίζω την κίνηση που αφήνει την ανθρωπιστική βοήθεια να περάσει. Ήταν μια πολύ επιφανειακή αντίδραση βέβαια μετά από την υπεραντίδραση στα όσα συνέβησαν πρέπει να δούμε αν η Χαμάς εισάγει όπλα στα παλαιστινιακά εδάφη, λόγω της χαλάρωσης του αποκλεισμού, τι θα συμβεί. Πρέπει αυτό να το προβλέψουμε. Την ίδια μέρα που δύο υπουργοί DUP ε, παρετήθηκαν από την ε, διοίκηση της Βόρειας Ιρλανδίας, εγώ περπατούσα γύρω τους καθώς στέκονταν στην κεντρική πλατεία κάνοντας τις, τις ε, συνεντεύξεις τύπου και πήγα να τους πω ποια ήταν η εμπειρία μου ως Προέδρου του Ιρλανδικού Κοινοβουλίου στην Επιτροπή Ευρωπαϊκή και καθώς έμπαινα ένας πολύ προφανής, προφανές τέλεχος, επιφανές μάλλον τέλεχος, είπε ότι δεν θα πάει, πρέπει να διαμαρτυρηθούμε με το Συνφέιν και η μόνη λύση θα είναι όταν θα υπάρξει το Ευρωπαϊκό Συνφέιν. Και αυτά ήταν τα δυο άκρα Μπορώ να σας πω ένα σωρό φορές για με τα πράγματα που είπαν όλοι ε, κατά τη διάρκεια όλων αυτών των ετών. Πρέπει να είμαστε δίκοι, λογικοί και ισορροπημένοι. Θέλουμε να προσπαθήσουμε να ανακουφίσουμε τον κόσμο και να καθοδηγούμαστε από το γεγονός ότι 800.000 από το 1,5 εκατομμύριο είναι κάτω από το 18. Τι θα φυθεί στην νέα γενεά, στην επόμενη γενεά, αν αυτή η υπόθεση συνεχιστεί. Ξέρω πως υπάρχουν προβλήματα με την πολιτική επικισμό, δεν ξέρω πώς αυτό θα αντιμετωπιστεί, αλλά ιδιωτικά κατεδίαν μου λένε πως μια λύση είναι πολύ δύσκολη, πρέπει να, να, ε, ε, δούμε και ποιος είναι ο ρόλος του Ιράν. Συνέβη και στην Ιρλανδία αυτό. Η Λιβύα έστειλε τότε η Λιβύη έστειλε τότε όπλα στον ε, IRA και ίσως και αλλού. Λοιπόν, Υπάρχουν, υπάρχουν άλλοι που χρησιμοποιούν την κατάσταση προς δικό του όφελο. Εγώ καλωσορίζω το γεγονός ότι ο κύριος Γκίνγκ θα έρθει. Αυτό ο άνθρωπο δεν φοβάται να μιλήσει όσον αφορά τα ανθρωπιστικά θέματα και επίσης καλωσορίζω το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργό Φαγιάντε θα έρθει να μας μιλήσει. Ευχαριστώ, ευχαριστώ εσάς και την αποστολή για την δουλειά που κάνατε εκεί και για την έκθεσή σας. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Κυρίως θα πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα στην ανθρωπιστική βοήθεια και μετά να δούμε μια ισορροπημένη προσέγγιση για τα πολιτικά θέματα. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you. Κυρία Πρόεδρε, πρωτού έρθω στην εκθεσή σας, Ελπίζω ότι ο φίλος και συνάδελφος Γκέι Μίτσελ ότι η έκθεση που δόθηκε για τον φόνο 16 ατόμων στη Βόρεια Ιρλανδία μπορεί να χρειάστηκε 38 χρόνια για να γίνει πραγματικότητα, αλλά τελικά έλαβε χώρα αυτή η έκθεση. Ζητώ συγγνώμη που δεν ήμουν παρόν για τη συζήτησή σα Υπήρχαν ορισμένοι καλεσμένοι από τη Σρι που συνόδευα. Αναρωτιέμαι, κυρία Πρόεδρε, αν αναμειχθήκαμε σε μια κατάσταση που δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε τα δέντρα από το δάσος. Σε άλλα μέρη του κόσμου, όταν υπάρχει μια ανθρωπιστική κρίση, την αντιμετωπίζουμε σαν ανθρωπιστική κρίση. Δεν αναμειγνύουμε την πολιτική με την ανθρωπιστική αυτή κρίση για τα περισσότερα μέρη του κόσμου. Το Σουδάν, παραδείγματος χάρη, ανεξάρτητα από τα καλά ή τα κακά του πρόεδρου Μπασίρ και τα λοιπά, εμείς δίνουμε ανθρωπιστική βοήθεια στο Σουδάν. Στη συγκεκριμένη αυτή την περίπτωση φαίνεται ότι έχουμε εμπλακεί στην πολιτική πτυχή των σχέσεων μεταξύ της Ισραηλινής κυβέρνησης και της Παλαιστινιακής Αρχής. Επομένως, απλοί άνθρωποι στην Παλαιστίνη έχουν υποφέρει η μεγαλύτερη μας δύναμη είναι ότι όταν θέλουμε να δώσουμε ανθρωπιστική βοήθεια, αποχωρίζουμε τα θέματα τα ανθρωπιστικά από τις πολιτικές θεωρήσεις. Μήπως θα πρέπει να ξαναγυρίσουμε και να δούμε την, επίτρο, την Επίτροπό μας για τα ανθρωπιστικά θέματα και να τη ζητήσουμε να κάνει μια έκκληση στη διεθνή κοινότητα και στο Ισραήλ να ασχοληθούν μόνο με τις ανθρωπιστικές πτυχές. Βέβαια, πρέπει να υπάρξουν διασφαλίσει, αλλά πρέπει να υπάρξει μια ανθρωπιστική αποστολή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, από ό,τι υπολογίζω, τα τελευταία δέκα χρόνια έχει δώσει περίπου 2 δισεκατομμύρια ευρώ στους, ε, για να αντιμετωπίσει την κρίση στην Παλαιστίνη. Αλλά δεν βλέπω να υπάρχουν τέτοιου είδους χρηματοδοτήσεις από τις αραβικές χώρες για ανθρωπιστικούς σκοπούς. Ίσως αυτό μπορούμε να κάνουμε και αυτό το υποβάλλω στην κρίση σας Ίσως θα πρέπει να διαχωρίσουμε την ανθρωπιστική προσέγγιση και πρωτοβουλίες από τις πολιτικές αντιμετωπίσεις και να πείσουμε τους συνομιλητές και από τις δύο πλευρές, τους Ισραηλινούς και τους Παλαιστινίους να εστιάσουν χωριστά στα δύο αυτά πράγματα. Ο κύριος Ντερόσα έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την έκθεσή σας και συγγνώμη που άρχισα γιατί ήμουν σε μια άλλη συνάντηση και καθυστέρησα. Εγώ ήμουν μέλος της ε, αντιπροσωπείας αυτής ως ε, πρόεδρος αντιπροσωπείας για την Παλαιστίνη. Θέλω να εκφράσω τη λύπη μου για το γεγονός ότι κάποια μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αποσύρθηκαν από αυτή την αποστολή θεωρώντας ότι ήταν μια αποστολή προπαγάνδας κατά του Ισραήλ. Αυτά είπε και ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, που φυσικά τελικά ήταν πάρα πολύ μακριά από την πραγματικότητα. Ποτέ δεν ήταν πρόθεσή μας να, κάνει, να κάνουμε κάτι τέτοιο. Λυπάμαι γι' αυτό που είχε σαν αποτέλεσμα και εγώ και ο Μπάσιαν Μπέλτερ που είναι ο πρόεδρος της αντιπροσωπείας με ε, ε, ο Μπάσιαν Μπέλτερ που είναι το για το Ισραήλ αποσύρθηκε από την αποστολή, κάτι το οποίο κατά την άποψή μου ήταν λαθασμένο. Νομίζω ότι αυτή η αποστολή ήταν πολύ θετική γιατί μας επέτρεψε να δούμε επιτοπίως τι ακριβώς λαμβάνει η χώρα χωρίς να χρειάζεται να βασιζόμαστε σε τρίτους. Χαίρομαι πολύ που ήταν μια αντιπροσωπεία τριών επιτροπών, προπολογισμών, εξωτερικών και ανάπτυξης και υπήρχαν οι πρόεδροι των δύο αντιπροσωπιών με το Ισραήλ και με την Παλαιστίνη. Αυτά δείχνουν λοιπόν τη σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όχι μονάχα τις ανθρωπιστικές πτυχές αλλά και τις πολιτικές πτυχές που αν θέλετε να κατηγοροποιήσετε τα θέματα αυτά ήταν αυτά τα οποία αφορούσαν και την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και τη δική μας Επιτροπή. Το πρόβλημα είναι ότι υπάρχει μια μεγάλη ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα, όχι σαν αποτέλεσμα φυσικής καταστροφής, αλλά λόγω πολιτικών αποφάσεων. Δεν είναι μια ανθρωπιστική κρίση όπως αυτή της ΑΕΤΗΣ. Είναι το αποτέλεσμα πολιτικών αποφάσεων. Και δεν είναι η μόνη κατάσταση εκτάκτου ανάγκης η οποία επισυμβαίνει στην περιοχή αυτή. Υπάρχει και πρόβλημα λειψιδρίας, όχι μονάχα στην Γάζα, αλλά και σε ορισμένε περιοχές στη Δυτική Όχθη. Οι Παλαιστίνοι δεν έχουν επαρκή πρόσβαση στο νερό, στις περιοχές τους. Τα ανθρώπινα δικαιώματα, για να το πω επίοικος, εμποδίζεται να ασκηθούν από τον τρόπο με τον οποίο το Ισραήλ διαχειρίζεται και διοικεί την Δυτική Όχθη. Η Παλαιστινιακή Αρχή έχει ένα έλεγχο μόναχα 40% του εδάφους της Δυτικής Όχθης. Τα άλλα 60% ελέγχονται από το Ισραήλ ή πλήρως ή από κοινού με την Παλαιστινιακή Αρχή. Και η κοιλάδα, στην κοιλάδα του Ιορδάνη η περιοχή ΣΥ ελέγχεται απόλυτα σαν στρατιωτική ζώνη από το Ισραήλ. Η δυνατότητα λοιπόν των Παλαιστινίων να διακινηθούν μέσα στη Δυτική Όχθη περιορίζεται τα μάλα και επομένως αυτό περιορίζει και τη δυνατότητα οικονομικής ανάπτυξης σε αυτή την περιοχή. Αν πάρετε την αναπτυξία, αν βγάλετε την αναπτυξιακή βοήθεια και τη βοήθεια που δίδεται για τη δημιουργία θεσμών στη Δυτική Όχθη, δεν θα υπήρχε καμία απολύτω οικονομική δραστηριότητα και ανάπτυξη στη Δυτική Όχθη. Όλα αυτά τροφοδοτούνται από τη δική μα βοήθεια. Είναι λοιπόν πάρα, ήταν πολύ σημαντικό και για την Επιτροπή Ανάπτυξη και την Επιτροπή Προπολογισμών να το δουν με τα ίδια του τα μάτια αυτή την κατάσταση. Εγώ πηγαίνω στην περιοχή αυτή δύο ή τρει φορέ το χρόνο και όπω είπε και ο συναδελφό μου, εγώ ε, απογοητεύτηκα για το γεγονό ότι κανεί από την Κνεσέτ εκτό από αυτού του δύο που αναφέρθηκαν δεν ήθελε να είναι παρόν. Δεν ήταν δυνατόν να έχουμε μονάχα δύο που θα μπορούσε να που θα μπορούσαν να είναι παρόντε για να αντιμετωπίσουν του εκπροσώπου τριών επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτό ήταν πραγματικό κρίμα. Συναντήσαμε τον αναπληρωτή Πρωθυπουργό και τον αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών. Είχαμε μια ειλικρινή συζήτηση μαζί του, όπω και με τον Σαλάμ Φαγιάτ και από μέλη του Κοινοβουλίου τη Παλαιστινιακή Αρχή. Θέσαμε το θέμα του Γκίλατ Σαλίτ και τη απελευθέρωσή του και άλλα θέματα επίση. Ήταν λοιπόν, κατά την άποψή μου, μια ευρέω χαρακτήρα ε, συζήτηση με την αντιπροσωπεία μα που είχε ε, ένα ευρύ χαρακτήρα και πιστεύω ότι αυτό θα πρέπει να είναι ο τρόπο με τον οποίο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να αντιμετωπίσει το θέμα αυτό στο μέλλον. Και θέλω να υπενθυμίσω ότι σήμερα την Τετάρτη το βράδυ στι 7 λαμβάνει χώρα μια συνάντηση της Υποεπιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που ακούει, θα ακούσει τις απόψεις ενός φορέα ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ισραήλ για την πίεση που ασκείται από τις αρχές του Ισραήλ στις μη κυβερνητικέ ε, οργανώσεις, ιδίως αυτές που ασχολούνται με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και από ό,τι κατανοώ θα είναι παρούσα και η πρεσβεία του Ισραήλ. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το παρακολουθήσουν τα μέλη της Επιτροπής μας και να δουν τι γίνεται. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας Άραβο-Ισραηλινός που είναι μέλος της Κνεσέτ, ο... η οποία κινδυνεύει να χάσει τα κοινοβουλευτικά της προνόμια γιατί συμμετέσχε στο στόλο αυτό που προσπάθησε να πάει στη Γάζα. Νομίζω ότι δεν μπορούμε να παριστάνουμε ότι μπορεί να αντιμετωπιστεί το θέμα αυτό δυστυχώς με το να μιλάμε μονάχα ιδιωτικά και ανεπίσημα με το Ισραήλ. Αυτή τη στιγμή δεν θα υπήρχε καν το, η χαλάρωση του αποκλεισμού αν δεν υπήρχε αυτή η εξέγεση της διεθνούς κοινή γνώμης. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι δεν αρκεί μονάχα να περνάμε ψηφίσματα όπως κάναμε την προηγούμενη εβδομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά θα πρέπει να δράσουμε επί τη βάση αυτών των ψηφισμάτων και θα πρότεινα η παράγραφος 10 που ζητάει μια αναδιάταξη της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Μέση Ανατολή θα πρέπει να τύχει συνέχεια και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να παίξει ηγετικό ρόλο για να τροποποιηθεί αυτή η πολιτική όχι μόνο για το συμφέρον των Παλαιστινίων αλλά και για τον ίδιο το συμφέρον των Ισραηλινών. Κύριε Σουνίμπερ, έχει το λόγο κυρία Πρόεδρε. Καταρχήν θέλω να σας ευχαριστήσω εκ βάθους καρδίας για την εκθέσή σας που έκανε σαφές το πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση σε αυτή την περιοχή του κόσμου. Όπως ελέγχθη εδώ δεν πρόκειται μονάχα για μια ανθρωπιστική κρίση. Και το λέω αυτό και από τη γερμανική οπτική γωνία γιατί εμείς έχουμε να αντιμετωπίσουμε και ένα ιδιαίτερο τραύμα ιστορικό. Ένα τραύμα το οποίο δεν πρέπει εμείς να το ενισχύσουμε με περαιτέρω ε, προκλήσεις, αλλά που θα πρέπει να μας οδηγήσει να έχουμε περισσότερη κατανόηση για όλα αυτά που έχουν ζήσει τα άτομα και από τις δύο πλευρές και για το γεγονός ότι η κατάστασή τους είναι πάρα πολύ δύσκολη. Νομίζω ότι το καθήκον μα αυτή τη στιγμή είναι να μην ενισχύσουμε του εξτρεμιστέ που υπάρχουν και από τι δύο πλευρέ, αλλά να υποστηρίξουμε αυτού οι οποίοι, του πολιτικού και του ανθρώπου που υποστηρίζουν μια πιο εξισορροπημένη πολιτική. Δεν θα πρέπει να σπρώξουμε το Ισραήλ στη γωνία, να το βάλουμε σε μια θέση από την οποία δεν θα μπορεί να ξαναβγεί. Θα πρέπει να κρατήσουμε πόρτες ανοιχτές για διάλογο και το γεγονός ότι τόσο λίγοι βουλευτές της Κνεσέτ ήταν έτοιμοι για διάλογο θα πρέπει να είναι ένας κόδωνας κινδύνου. Θα πρέπει να μας δείξει ότι δεν έχουμε δημιουργήσει αρκετή εμπιστοσύνη. Και πρέπει να υπάρχει εμπιστοσύνη και από τι δύο πλευρέ, όχι μονάχα από τη μία. Θα πρέπει να ενισχύσουμε την εμπιστοσύνη και των δύο πλευρών, γιατί αυτό ο διάλογο είναι κάτι το οποίο το απαιτούμε. Είναι ο μόνο δρόμο μέσα από τον οποίο μπορούμε να βοηθήσουμε του ανθρώπου τη περιοχή να ξεπεράσουν τα προβλήματα αυτά. Γι' αυτό έλαβα το λόγο και εγώ. Θεωρώ ότι είναι δύσκολο να μιλάμε για προσκλήσεις μόνο της μίας πλευράς. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να έχουμε επαφή και με τους δύο εταίρους και με τις δύο πλευρές να έχουμε μια ισορροπία. Να έχουμε ή δυνατόν προσκλήσεις εκπροσώπων και από τις δύο πλευρές. Πολύ σύντομα, Πρόεδρε, δύο λέξεις. Καταρχήν πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό, όπως είπα, για τις ανθρωπιστικές ε, ανάγκες και το έχω πει ε, στο Κοινοβούλιο πριν και μετά τα περασμένα Χριστούγεννα και πιο πρόσφατα και το επαναλαμβάνω για να σημειωθεί στα πρακτικά. Και επίσης, ε, αν πίστευα ότι η, ότι η συγνώμη του Πρωθυπουργού ήταν αρκετή, ναι, ήταν πολύ ευπρόσδεκτη και σίγουρα τέτοια βήματα μας πάνε μπροστά. Καλώς. Ευχαριστώ όλους σας για τα ερωτήματα, για τη συμβολή σας. Έχουν δειχτεί πάρα πολλά θέματα. Και ειλικρινά δεν είναι δυνατό να έχει κανείς, να εύκολα να οδηγηθεί σε μια κατάληξη. Για μένα όμως έφτασε το σημείο για τον καθένα να ξεφύγει από κλισέ, να επαναβάνει κανείς ό,τι λέγεται εδώ και 60 χρόνια, να δούμε πλέον την πραγματικότητα στα μάτια. Οι εκπρόσωποι του ΚΝΕΣΕΤ θα μπορούσαν να δεχθούμε εμάς τους εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εκπροσωπούμε 500 ε, εκατομμύρια ε, κόσμο εμείς θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι το ότι αρνήθηκε σε εμά το, το το διάλογο αυτό δείχνει κάτι. Θα πρέπει και εμείς να καταλάβουμε όμως ποια είναι η κατάσταση στο Ισραήλ, πού ακριβώς, πώς μπλοκάρεται έτσι το Ισραήλ, πώς έχει καταλήξει σε μια απομονωμένη κατάσταση να κλείνεται έτσι σαν χώρα για μας που είμαστε μέλος του κουαρτέτου, που είμαστε δωρητές, δείχνει ότι κάτι δεν πάει καλά. Ότι δεν υπάρχει δυνατότητα κατανόησης. Ότι οικοδομήσαν ένα κράτος ε, σε αντιπαράθεση με τον υπόλοιπο κόσμο και πραγματικά τα πράγματα έχουν πάρει μια τέτοια διάσταση που εμείς σαν υπεύθυνα άτομα, πολιτικά όντα, θα πρέπει να πούμε ότι είναι τρέλα. Και όπως λέει εδώ ο συνάδελφός μου, ε, για, για το θέμα της ανθρωπιστικής βοήθειας να υπάρχει μια ένα διαχωρισμός. Εγώ θα ήθελα να πω ότι έχουμε να κάνουμε ένα θέμα το οποίο κρατά 63 χρόνια, θα πρέπει να αναλάβουμε τις ευθύνε μας, να δούμε ποιε είναι οι δυνατές λύσεις, ποιε είναι οι σωστέ λύσεις. Και ευχαριστώ τον κύριο Μισελ που ανέφερε εδώ πέρα τις προσωπικές του ε, μνήμες, αναφερόμενος στην Ιρλανδία. Πραγματικά έχει μια εμπειρία και ειλικρινά αυτός ανάμεσά μας είναι αυτός που έχει μια ανάλογη εμπειρία, την πιο σωστή εμπειρία. Θεωρώ ότι κατά κάποιο τρόπο ε, η περίοδος κατά την οποία η Ευρώπη ήταν σιωπηλή και το ότι αισθάνεται και μια ανοχή, αυτή η περίοδος πρέπει να κλείσει. Και όταν έχουμε να κάνουμε μια κατάσταση ότι δεν γίνονται σεβαστά ψηφίσματα εδώ και τόσα χρόνια, βλέπουμε ότι οδηγείται κανείς σε μια κατάσταση όπου η αριστερά δεν γνωρίζει τι πει η δεξιά. Απ' τη μια έχουμε επικισμούς και απ' την άλλη διαπραγματεύσεις. Έφτασε λοιπόν η στιγμή για την Ευρώπη. Ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, ούτω ώστε όχι μόνο να είναι ε, παθητικός εταίρος, αλλά να πάρει μια ε, σωστή θέση στη διπλωματία και να επιβάλλει μαζί με άλλους εταίρους μία λύση. Και όντως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να πάρει τη θέση του να απαιτήσει από την ε, είπα το πρόσωπο να παρουσιάσει ένα πρόγραμμα δράσης μαζί με όλα τα μέσα που έχουμε, με όλα τα πολλά που έχουμε στη διάθεσή μας. Και πραγματικά υπολογίζω στη συνοχή της ομάδας μας και λυπάμαι που το ΣΕΡ δεν έλαβε... Δεν συμμετείχε στις διαπραγματεύσει. διαπραγματεύσεις. Έχουμε το όνομα Μλάγιος Μπόκρος. Και είναι ένα άτομο το οποίο συμμερίζεται τις απόψεις μας. Έκανε ακριβώς την ίδια ανάλυση με μας και είχε πραγματικά, ήταν πολύ αυστηρός, επικριτικός και επιθυμούσε να συνεργαστεί με την ομάδα μας. Και ελέγχθη ότι είμαστε όλοι ενωμένοι μαζί να δουλέψουμε για να οδηγηθούμε σε μια σωστή έκβαση. Ευχαριστώ. Alors, donc... Λοιπόν, ε, εξαντλήσαμε από ό,τι φαίνεται την ημερήσια διάταξή μας. Σας υπενθυμίζω αύριο το πρωί ξεκινάμε με τους συντονιστές στις ε, 9, 9 και θα ξαναρχίσουμε 10 και 4 τη συνεδρίαση. Τίποτα άλλο για απόψε αύριο στις 10 και 4. 9 οι συντονιστές. Ευχαριστώ.